Okay, colleagues and uh, friends, perhaps we can look to uh, make a start. Καλώς ε, συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε αφού είναι ήδη 3 και 5. Ε, όπως θα είδατε δεν είναι εδώ μαζί μας η πρόεδρος ε, Γκρέσλε, οπότε δυστυχώς ε, ε, αστεύεται ο πρόεδρος, θα έχετε να κάνετε μαζί μου για το υπόλοιπο της απογευματινής μας συνεδρίασης. Όπως θα είδατε, έχουμε μία σειρά από θέματα στην μέσα διαταξή μα και σημαντικέ συζητήσει. Οπότε για κάθε ένα από τα σημεία που θα συζητήσουμε έχουμε μόνο μισή ώρα. Οπότε θα ήθελα οι συνάδελφοι να τηρήσουν τους χρόνους αγορευσή τους και να είναι όσο το δυνατόν συντομότεροι. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο σημείο είναι η έγκρισή της. Δεν νομίζω πως υπάρχουν αντιρρήσεις ε, στην ημερήσια διάταξη, οπότε θεωρούμε πως εγκρίνεται. Επόμενο ε, σημείο είναι ανακοινώσεις του Προέδρου στα Cont News θα δείτε ποια allowances υπάρχουν διαθέσιμα και θα δείτε, και επίσης, ε, θα δείτε συγγνώμη, ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες και θα δείτε ότι έχουμε web streaming. Ε, και είμαι σίγουρος ότι έχουμε εκατομμύρια θεατές οι οποίοι είναι κολλημένοι στις οθόνες των υπολογιστών τους και μας παρακολουθούν. Τώρα, περνάμε στο σημείο 3 της σήμερα σας διάταξης, δηλαδή η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση της Επιτροπής των συμφωνιών εταιρική σχέση και των προγραμμάτων του 2014-2020 σχετικά με τη συνοχή και ούτω καθεξής. Το αρμόδιο μέλος του ελεκτικού συνεδρίου ε, ήταν ο κύριος Μπάρκος, οπότε θα του δώσουμε λίγα λεπτά για να κάνει την παρουσίαση του. Ε, έχετε το λόγο κύριε Μπάρκο. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ Πρόεδρε ε, και αξιότιμη κύριε Σιγητά Πυρίνστη και αξιότιμοι συνάδελφοι. Ε, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020 και όπου εξετάμε κατά πόσο διαπραγματεύτηκε αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα, ε, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν πιο αποτελεσματικά ή, ε, αυτά τα προγράμματα και οι συμφωνίες με τη στρατηγική του 2020. Και επίσης είχε στόχο να ε, αιτιολογηθούν οι ανάγκε επενδύσεων και τα αποτελέσματα και να τεθούν και προϋποθέσεις ό,τι αφορά την μέτρηση των ε, Επιτόσεων. Όπως είπα τώρα στον ε, κύριο Πυρίνσκι κατά την προπαρασκευαστική μας συνεδρίαση, αυτή η ε, πρώτη έκθεση θα συμπληρωθεί από μια σχετική έκθεση αργότερα φέτος σε ό,τι αφορά τις εκ των προτέρων ερεσιμότητες. Τώρα, οι εταιρικέ σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, σχέδια στρατηγικών επενδύσεων όπου τα κράτη-μέλη αναφέρουν τις ε, προτεραιότητες τους ό,τι αφορά τις δαπάνες τους από τα ε, ευρωπαϊκά διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία. Και έγινε διαπραγμάτευσή του το 2014 και η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε 387 επιχειρησιακά προγράμματα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνεχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συνολικά θεωρήσαμε πως ήταν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις ε, εταιρικές σχέσεις και τα επιχειρησιακά προγράμματα και ε, τηρήθηκαν οι κατάλληλε προθεσμίε και έγινε η κατάλληλη ευθυγράμμιση σε ό,τι αφορά ε, και του ε, στόχου τη ε, στρατηγική Ευρώπη 2020. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ε, η Επιτροπή να εναρμονίσει τις ε, ε, συμφωνίες σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική παρακολούθηση ανάμεσα στα ταμεία και, την, και να διασφαλίσει μια συνεκτική, ένα συνεκτικό ορισμό των δικτών επιδόσεων. Και αυτό βέβαια ήταν απαραίτητο ώστε να υπάρξει μια καλή άθρηση και σύγκριση των δεδομένων επιδόσεων μεταξύ των προγραμμάτων. Και επίσης επειδή υπάρχει ένας πολύ υψηλός αριθμός δικτών, υπάρχει ε, και ε, ο κίνδυνος ε, επιπρόσθετου δικηρικού άχθους. Τώρα, να, πω κάποια, να επιστρέψω κάποιε λεπτομέρειε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Το νομοθετικό λοιπόν πακέτο για την πολιτική συνοχή τη περίοδου 2014-2020 υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, δηλαδή πέντε μήνες αργότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη υπέβαλαν τι ε, συμφωνίε εταιρική σχέση εγκαίρω ε, και ε, κατά μέσο όρο η Επιτροπή τα υιοθέτησε εντό πέντε μηνών, δηλαδή ένα μήνα ταχύτερα, σε σύγκρουση με τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφορά στι προηγούμενε περίοδου. Επίση, Ήδη το 2012 η Επιτροπή ξεκίνησε τι άτυπε διαπραγματεύσει με τα κράτη-μέλη και ένα καινοτόμο στοιχείο ήταν το γεγονό ότι άρχισε να εκδίδει position papers, δηλαδή έγγραφα σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή τη, που περιείχαν ανάλυση των κυρίων προκλήσεων που αντιμετώπισε το κράτη, κάθε κράτο-μέλο σε ό,τι αφορά την πρόοδο ε, για την επίτευξη των ε, στόχων τη Ευρωπαϊκή 2020 και περιείχε και τι απόψει τη Επιτροπής σε ό,τι αφορά τι κυριότερες προτεραιότητε χρηματοδότηση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν υπέβαλαν τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα εγκαίρω και η Επιτροπή τα υιοθέτησε εντό των προβλεπόμενων ε, προθεσμιών του κανονισμού. Τώρα, οι διαπραγματεύσει επί των επιχειρησιακών προγραμμάτων μεταξύ Επιτροπή και κρατών μελών ήταν πιο δύσκολε. και ε, κύριο λόγοι ήταν ότι υπήρχαν επιπρόσθετε ε, ε, για παράδειγμα εκ των προτέρων ευσημότητε ή η συγκεκριμένη απέτηση να υπάρχει πιο συγκεκριμένη λογική των παρεμβάσεων, να υπάρχει έκθεση των, προγραμμάτων, ε, ε, των προβλημάτων μηχανοργάνωσης, αναφορά διαφόρων αιτιολογήσεων σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις από την Επιτροπή και ούτω καθεξής. Με βάση λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις, εμείς συνιστούμε η Επιτροπή να υπαρχει πιο συγκεκριμενη λογικη των παρεμβασεων να υπαρχει εκθεση των των προβληματων μηχανογάνωση, αναφορα διαφορων αιτιολογησεων σε οτι αφορα τι εγκρισει απο την επιτροπη και ουτω καθεξης με βαση λοιπον αυτέ τι παρατηρήσει, εμεί συνιστουμε η επιτροπη να παρουσιασει εγκαίρω ε, τι νομοθετικέ τη προτάσει ό,τι αφορά την ε, πολιτική συνοχή για την περίοδο μετά το 2020, έτσι ώστε να υπάρχει ο κατάλληλο χρόνο για τι νομοθετικέ αρχέ να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει και να ολοκληρώσουν τι διαπραγματεύσει. Τέλο, ε, μάλλον δεύτερον, σε ό,τι αφορά την τις δαπάνες στον τομέα της συνοχής και τις προτεραιότητες του 2020, θεωρήσαμε πως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να οριοθετηθεί η χρηματοδότηση των επενδυτικών και διαθωτικών ταμείων σε ό,τι αφορά τις ε, προτεραιότητες ε, επενδύσεων στον τομέα της ε, στρατηγικής συνοχής. Τώρα, οι απαιτήσει σε ό,τι αφορά την εστίαση σε θεματικά ζητήματα πληρώθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη την ε, επίτευξη των στρατηγικών αποτελεσμάτων και τα επιπρόσθετα κανονιστικά μέτρα και τις διαθωτικές μεταρρυθμίσεις ε, σημειώσαμε ότι η Επιτροπή αξιοποιεί όλο ένα και περισσότερα ε, τον προγραμματισμό των κονδυλίων των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ώστε να ε, επηρεάζει περισσότερο την οικονομική διακυβέρνηση από την πλευρά των κρατών μελών. Επίση, σε ό,τι αφορά τα περισσότερα από τα προγράμματα που εξετάσαμε, υπήρχε μια πιο συνεκτική λογική επανέμβαση. Ωστόσο, μερικέ φορέ οι σχετικέ πληροφορίε δεν είναι τόσο συνεκτικέ και ε, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη που αξιοποιούν παρεκκλήσει ή οικονομικέ πληροφορίε οι δημοσιονομικές πληροφορίες των προγραμμάτων δεν επιτρέπουν να ε, ε, επαληθευτεί κατά πόσο αυτή η εστίαση στους θεματικούς τομείς τελικά πληρείται ή όχι. Με βάση λοιπόν αυτές τις ε, παρατηρήσεις εμείς συστούμε στα κράτη-μέλη να παρέχουν τις δημοσιονομικές πληροφορίες στην Επιτροπή που αυτή χρειάζεται ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με την την εστίαση στις κυρίες προτεραιότητες. Επίσης, μια σχετική σύσταση προς την Επιτροπή είναι να διασφαλίζει ε, την εστίαση των ε, κονδυλίων των ε, διευθυντικών και επενδυτικών ταμείων στους κύριους θεματικούς στόχους, όπως έχουν από τα κράτη-μέλη. Ε, τώρα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο σημαντικότερο πρόγραμμα, δηλαδή τον περίπλοκο χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων τη περίοδου 2014-2020, που αποτελεί και βέβαια τη συνέπεια μια σειρά από παράγοντε. Δηλαδή, ο αριθμό των αξώνων προτεραιότητα στα κράτη-μέλη, ο αριθμό των προτεραιοτήτων επενδύσεων, αλλά και ο αριθμό των κατηγοριών των περιοχών. Και εδώ σα καλώ να ρίξετε μια ματιά στον ε, τρισδιάστατο πίνακα που περιλαμβάνεται εκεί στην, ε, στο κυκλικό διάγραμμα, στο παράδειγμα 3 στην σελίδα 89 της έκθεσής μας. Αν λήξετε λοιπόν εκεί μια ματιά θα δείτε ότι πραγματικά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλούστευση. Χρειάζεται περαιτέρω απλούστευση σε όλα τα επίπεδα. Ε, πέραν αυτού η μουσιονική παρακολούθηση των ε, ε, επενδύσεων διαφέρει μεταξύ του Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Για το ERDF δηλαδή, η σχέση μεταξύ των δράσεων και της χρηματοδότησης δεν μπορεί να καθοριστεί με, με ευκολία, γιατί ακριβώς οι δημοσιονομικές πληροφορίες δεν αντιστοιχούν στις προτεραιότητες των επενδύσεων. Ενώ σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο υπάρχει αυτή η ευθυγράμμιση. Ε, ταυτόχρονα, ε, στο ERDF το, ο ίδιος τομέας ε, παρέμβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ό,τι αφορά διαφορετικούς θεματικούς ε, στόχους. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της προόδου γιατί δεν γνωρίζουμε τελικά πόσα κονδύλια επενδύονται σε ό,τι αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών προτεραιοτήτων επενδύσεων. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα και τις διαφορές μεταξύ RDF και ESF και τις σχετικές προσεγγίσεις, σας καλώ να ρίξετε μια ματιά ε, στο διάγραμμα που έχουμε ε, υπαριθμό 15 σελίδα 74, γιατί καταδεικνύει ακριβώς πολύ ότι έχουμε πολλές, πολλά, πιο, πολλά πλεονεκτήματα, αν θέλετε, ισχυρά σημεία σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο σε σύγκριση με το RDF και το αντίθετο. Τώρα, έχουμε και κοινού δείκτε οι οποίοι υπάρχουν μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο. Δηλαδή πάρα πολλοί, 2.955 για το ERDF και 1.976 για το ESF. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ε, έχουμε ακόμα ε, μεγαλύτερο αριθμό, ακόμα πιο περίπλοκο, ακόμα πιο περίπλοκα δεδομένα και δυσκολίες σε ό,τι αφορά μια ασόρευση των σχετικών δεδομένων που να έχει νόημα. Ε, επίσης δεν υπάρχει ένας κοινό ορισμός των outputs, των αποτελεσμάτων σε αυτού αν θέλετε αριθμού και των results, των αποτελεσμάτων, γενικών αποτελεσμάτων. Ε, και τα αποτελέσματα του ESF ε, ε, αναφέρονται σε τα αποτελέσματα των πανεβάσεων σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντε ή του φορεί οι οποίοι λαμβάνουν υποστήριξη. Ενώ σε ό,τι αφορά το ERDF έχουμε να κάνουμε με μάκρο διαστάσεις ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις επενδύσεις οι οποίες υποστηρίζονται. Ε, Παρ' όλα αυτά θεωρούμε πως θα μπορούσαν να υπάρχουν καλύτερα δεδομένα επιδόσεων σε ό,τι αφορά τα outputs, δηλαδή τα αποτελέσματα σε απόλυτους αριθμούς, έτσι ώστε να υπάρχει ένας προϋπολογισμός στο μέλλον για την περίοδο μετά το 2020 που θα, θα προσανατολίζεται περισσότερο στις επιδόσεις. Με βάση λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις προτείνουμε στην Επιτροπή να υπάρχει μια κοινή ορολογία στο μέλλον σε ό,τι αφορά outputs και results και να προταθεί αυτή η ορολογία να συμπεριληφθεί ληφθεί στο δημοσιονομικό κανονισμό και να ακολουθούνται αυτοί οι ορισμοί για την περίοδο μετά το 2020. Επίση, θα πρέπει να γίνει και μία ανάλυση σε ό,τι αφορά τα προγράμματα τη περίοδου 2014-2020 και να ε, ε, καθοριστούν και συγκεκριμένοι δείκτε οι οποίοι είναι οι πλέον συναφεί σε ό,τι αφορά τα output και αυτοί να ληφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά ε, την αξιολόγηση του αντικτύπου των παρεμβάσεων των κρατών μελών. Θα πρέπει να σταματήσει δηλαδή η χρήση δικτών οι οποίοι είναι Περί τι. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν τροποποίησει των σχετικών προγραμμάτων στο πλαίσιο τη ίδια ε, περίοδου προγραμματισμού. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των προγραμμάτων, όπω φάνηκε στι ταξιολογήσει, αυτό ε, συνεχίζει να ισχύει. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτούμενε δράσεις και τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται και συστηματικά από τα κράτη-μέλη και να αφαίρονται στην ε, Επιτροπή. Ωστόσο, οι δείκτε αποτελεσμάτων του ERDF δεν απηχούν τα άμεσα αποτελέσματα των ε, προγραμμάτων και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα εκτός και αν τα κράτη-μέλη ε, ξεκινούν να συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα συμπληρωματικά. Τα εν λόγω δεδομένα ούτως ή άλλως δεν υποβάλλονται σε συμπληρωματικές ε, εκθέσεις και εξέταση. Οπότε συνιστούμε στην Επιτροπή να διαδώσει, να χορηγήσει στα κράτη-μέλη καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις προκειμένου να αξιολογούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο αντίκτυπος, η των και να υποστηρίζει η Επιτροπή τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση των ε, σχεδίων αξιολόγησή του. Τέλο, ε, θεωρούμε πω οι διαφορετικέ απαιτήσει σε ό,τι αφορά του κανονισμού ε, για το κάθε ταμείο και σε ό,τι αφορά και την συλλογή των δεδομένων επιδόσεων σε σχέση με outputs και results, όπω σα ανέφερα μόλι τώρα, αποτελεί μια σημαντική αδυναμία μέσα στο σύστημα. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα παρακολούθηση σε ό,τι αφορά την ε, συγκεκριμένου δείκτε επιδόσεων και θα πρέπει να λάβουν υπόψη του ε, συγκεκριμένε ε, μεθοδολογίε και να μην υπάρχει πλέον ένα υπερβολικό αριθμό δείκτων. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει ένα πολύ υψηλό διοικητικό άκτο. Γι' αυτό λοιπόν συνιστούμε η κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που υπάρχουν στι αιτήσει εκθέσει εφαρμογή και τι αξιολογήσει, προκειμένου να προβαίνει σε συγκριτικέ αναλύσει και προκειμένου να υπάρξει ακριβώ η συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων προπαρασκευαστική δηλαδή για την περίοδο του ε, μετά το 2020 και όπου αυτό ε, ενδείκνεται θα πρέπει να ε, εφαρμόζεται και η προσέγγιση του performance budget, δηλαδή του προπολογισμού που προσανατολίζεται στις επιδόσεις για την περίοδο χρηματοδότησης μετά το 2020 στον τομέα της συνοχής, αξιοποιούντας τα δεδομένα με βάση τις της, κόστος μονάδες κόστους που χρησιμοποιούνταν στην τρέχουσα περίοδο. Κυρίε και κύριοι, λοιπόν, για να κλείσω την δική μου παρουσίαση, συνοψίζω ε, αναφέροντα και την, ε, τον τίτλο τη έκθεσή μα, ότι η Επιτροπή δηλαδή ήταν αποτελεσματική στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρική σχέση 2014-2020 και τα, σε ό,τι αφορά και τα προγράμματα για την καλύτερη στόχευση των, ε, των δαπανών σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του Europe 2020, αλλά υπάρχουν ολοένα και πιο ε, περίπλοκες ε, συμφωνίες σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη μέτρηση των επιδόσεων και αυτό δημιουργεί ανησυχία. Σας, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολλά για ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστούμε, ήταν πάρα πολύ ε, ολοκληρωμένη παρουσία σας και τώρα το λόγο ο κύριος Πυρίνσκι, ο εισηγητής μας και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή του Ελληνικού Συνεδρίου, τον κύριο ε, Βάλκο, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια κατά την εισήγηση. Είναι αλήθεια ότι έπιασε την ουσία αυτή της ε, ειδική έκτακτη έκθεσης. Συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση, γι' αυτό και το επόμενο θέμα, και αυτή για την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε το 7ο φόρουμ για την συνοχή, το οποίο ε, επίκειται και είναι βασικές ότι η πολιτική της συνοχής αναγνωρίζεται αφενός ως ε, το πιο σημαντικό μέσο επενδύσεων στην Ένωση, αλλά επίσης ε, πρόκειται να υποστεί και μίζωνα μεταρρύθμιση. Άρα να μην ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια πρόκληση να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή την πολιτική μετά το 2020 και να το κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Και τώρα για να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τις συστάσεις που επεσήμανε αυτή η εκτακτή έκθεση. Η ειδική έκθεση τέλος πάντων γιατί είναι τα ζητήματα τα οποία αφορούν την περίοδο 2020 και πρώτα-πρώτα. Το θέμα είναι ο σωστός χρονισμός. Το αν είμαστε έγκυροι. Να πρέπει να εξασφαλιστεί ακριβώ το ότι θα πρέπει οι νομοθετικέ προτάσει εγκαίρω να τυπώνται τόσο ώστε να υπάρχει περιθώριο για πραγματεύσει. Δεν ξέρουμε πριν το 2014 πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος, τι δυσκολίε είχαμε και βεβαίω υπάρχει πάντοτε σπάνια στους νευροτούς πόρου και πολλέ προκλήσει να αντιμετωπιστούν και προβλήματα να επιληθούν και επομένω είναι ξεκάθαρα υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με το άρθρο 25 του ε, κανονισμού του πολιετού πλαισίου ότι θα πρέπει πριν την 1η Ιανουαρίου του 2019 να έχουμε προχωρήσει αυτό το μέτωπο και όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή ότι θα κάνει κάποια πρόταση για νομοθετικά μέτρα στην συνέχεια. Αυτές οι επισημάνσεις νομίζω πρόεδρε αξίζουν προσεκτική αξιολόγηση. Έλεγε ότι αυτή η προθεσμία δεν θα τηρηθεί πλέον τη Κομισιόν για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ίσως πάμε για το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 18. Οπότε η πρόταση δεν θα έρθει αμέσω με την παρουσίαση του πλαισίου του δημοσιονομικού. Ε, θα έχει συνέπειες. Οπότε ερωτοξής απλό. Τι θέση παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι πιστεύει ότι θα γίνει μέχρι αλλά και μετά την 1η Ιανουαρίου, τι θα γίνει με το νομοθετικό πλαίσιο στην παράγραφο 4 δε του εγγράφου εργασίας το οποίο έχω ε, συντάξει υπάρχει ακριβώ αυτό το θέμα, και το φύγουμε ότι προς το κάνα, προς το κούμιο, ότι λέει θα παρουσιάσει αμέσως μετά, ε, αμέσως πριν την 1η 18, την πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ξεκάθαρη σύσταση του ελληνικού συνεδρίου, τι γίνεται δηλαδή με αυτό το τόσο σημαντικό νομοθετικό μέτρο που αφορά την ε, πολιτική συνοχή με το 2020. Επίση, το θέμα τι γίνεται στου θεματικού στόχου, τι γίνεται με τη θεματική συγκέντρωση. Αποδέχεται η Επιτροπή αυτή τη σύσταση, όμω και προκειμένου έχουμε κάποια ζητήματα. Διότι στην έκθεση κάτι αναφέρεται για κάποια ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2015 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την μεγιστοποίηση των, ε, της χρήσης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διαρθρωτικών και ε, διαρθρώσεων και επενδύσεων τέλο πάντων και το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε τι έγινε και με αυτό. Η ιδέα η Επιτροπή σε Ευέθυνση υπενθυμίζω ότι με συνένεση δήλωσε ότι εκπλήσεται με αυτά έχουμε απλώ αυτή την ανακοίνωση με κάποιο είδου στοιχεία για τι διαπραγματεύσει όσον αφορά τι εταιρικέ συμφωνίε και τα λειτουργικά προγράμματα, τα επιχειρησιακά προγράμματα. Άρα θα πρέπει να δούμε πώ συμβάλλουν αυτά τα ταμεία, τι αξιολόγηση έχει γίνει για το ρόλο του. Τι θέση παίρνει για θεματική σύγκρουση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης έχουμε τη σύσταση υπαριθμών 3 που αφορά την ορολογία και τους ορισμούς. Τι θα πει output και τι θα πει result. Δέχεται εν μέρη η Επιτροπή τη σύσταση. Και αναφέρει ότι το παρόντος δεν είναι στέση να προβεί σε κάποια δέσμευση όσον αφορά κάποια νομοθετική πρόταση για την περίοδο μετά το 2020. τώρα λέμε για συγκεκριμένους κανονισμούς αναφερετικού χαρακτήρα και εμείς έχουμε περάσει και από τις τριμερείς διαπραγματεύσεις αλλά θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι θα κάνει για αυτό το τόσο βασικό πρόβλημα με σαφήνεια να τοποθετηθεί για το τι θεωρεί ότι πάει να πει result και τι θα πει output. θεωρεί ότι λειτουργεί εύρυθμα η πολιτική συνοχή. Οι υπόλοιπε συστάσει 4 και 5 δεν δημιουργούν πρόβλημα στην Επιτροπή. Έχει αυτού του κοινού δείκτε για την ανάλυση όσον αφορά τη μελέτη των επιπτώσεων και η πέμπτη αναφέρει τις καλές πρακτικές το gold Τώρα για να δούμε τι γίνεται με την σύσταση παριθμών 6. Εδώ θα πρέπει να υιοθετήσει τη συγκριτική αξιολόγηση επιτροπή και να εφαρμόσει το performance budget ούτως ώστε να βελτιώσει το output σε σχέση με τις ε, Χρησιμοποιούμε ένας χρησιμοποιούμενους πόρους. Υπάρχουν πάντα και εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτά έχουν επισημαθεί και από το Κοινοβούλιο στο παρελθόν σε διάφορα ψηφίσματα. Γιατί εδώ υπάρχει το βασικό πρόβλημα του πώς αυτοί οι πόροι, αυτές οι επιστροφές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους στόχους, και πώς να τους πέτυχαν. Και ξέρουμε ότι η συγκυρία, το περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από δυσπιστία προς τις πολιτικές και τις ε, πολιτικές συνοχής. Υπάρχει ο λαϊκισμός που επηρεάζει και διαμορφώνει το σκέπτεστε των πολιτικών και των ηγετών. που είναι πάρα πολύ διστακτική και προσεκτική όσον αφορά τις πολιτικές συνοχές και τη διαμόρφωσή τους. Οπότε το θέμα είναι εδώ να δούμε συγκεκριμένα. Πώς αξιολογείται η πολιτική συνοχής, πέτυχε, αλλά αυτά να προκύψουν ξεκάθαρα. Τώρα έχω άλλε τρει σκέψει που ταυτόχρονα είναι προβληματισμό και σύσταση. Τι πάει να πει απλούστευση. Τι πάει να πει και έγινε. Δεν έγινε. Πρόσφατα. Γίνανε όλα μέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλεπόντουσαν, αλλά αυξήθηκε η πολυπλοκότητα. Και είπαμε ότι χρειάζονται και δυο και τρεις παραπάνω εκθέσεις για αυτό τον κύκλο άσκηση της πολιτικής συνοχής. Επομένως, η απλούστευση παραμένει ένα κατεπήγον ζητούμενο. Τώρα, σαν αφορά την προσβασιμότητα στους πόρους και κατά πόσο πρέπει αυτό να διευκολυνθεί, ακούσαμε τα σχετικά. πρέπει αυτό να μας απασχολήσει και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Επίσης θα πρέπει όλα αυτά να τα θεωρήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο μέσα στο οποίο να τα επιδιώξουμε γιατί είχαμε στο παρελθόν τα σχετικά με την περίοδο 2020 μέχρι τότε μάλλον αλλά τι θα γίνει μετά το 2020 το μέλλον άδειλο αυτό η αμηχανία φαίνεται από παντού Άρα χρειαζόμαστε κάποιο είδους ορόσημα, κάποιο είδους μπούσουλα. Περιμένουμε να μας διαφωτίσει και ο πρόεδρος Γιούγκερ το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την σε βάθος παρουσίαση. Έχετε υποβάλει και ορισμένες ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω τώρα που θα λάβει το λόγο να μπορεί να απαντήσει. Θα δώσω όμως το λόγο πρώτα στα μέλη. Νομίζω Μαρτίνα πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ βεβαίως και το ελεγκτικό συνέδριο και τον κύριο Πυρίνσκι για τα ενδιαφέροντα έγγραφα. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια του εισηγητού μας που περιγράφει και στο έγγραφο εργασίας του και τον ευχαριστώ. Τρία συγκεκριμένα σχόλια. Ανησυχώ και εγώ για την καθυστέρηση των πέντε μηνών όπως και εσείς και το συνέδριο. Δεν είναι καλό μήνυμα πρέπει να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένες έγκαιρα και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να δαπανηθούν σωστά οι πόροι χωρίς να επιταχύνουμε με περιττό τρόπο στο τέλος της περίοδου, δηλαδή να βιαζόμαστε. Πρέπει να διασφαλιστεί επίσης ώστε όλα, όλες οι εταιρικέ συμφωνίες να εγκριθούν έγκαιρα και πάντως έγκαιρα ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν και τα λειτουργικά προγράμματα πριν από την επόμενη περίοδο προγραμματισμού γιατί οι καθυστερήσεις φέρνουν μια την άλλη. Και επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα σε όλες τις προγραμματικές περιόδους. Θα πρέπει να μπορούν να αρχίσουν και ανεπίσημες οι διαπραγματεύσει με τις χώρες μέλη πριν μάλιστα από την περίοδο για να φανεί και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι οι Κομισιόν ή και χώρες μέλη δεν έχουν διδαχθεί από το παρελθόν διότι βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τα ίδια σφάλματα, δηλαδή καθυστερημένη έγκριση επιχειρηματικών προγραμμάτων, καθυστερημένη απορρόφηση, ε, λιγότερη χρήση ε, των ε, ταμείων μετά από τις μάλιστα μετά από τις προγραμματικές περιόδους, μετά την εκνοή τους δηλαδή, πρέπει να διδαχτούμε από τα σφάλματα του παρελθόντος. Και αυτό είναι ένα θέμα νομίζω το οποίο θα πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο, ανησυχώ για τις χιλιάδες performance indicators που δημιουργούν οι χώρες μέλη και οι κοινοί δείκτες τελικώς ξεπερνιούνται σε αριθμό από, τα, από τους ειδικούς δείκτες, ειδικούς προγραμματικούς δείκτες. Χρειάζεται συγκεκριμένο αριθμό δικτών και αυτό το επιβεβαιώνει και το ελεγκτικό συνέδριο στην ανάλυση του, γιατί αυτά αλλιώ θα οδηγήσουν σε έξτρα διοικητική επιβάρυνση και θα ήθελα να παρακαλέσω να ρωτήσω μάλλον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ακριβώ βρίσκεται σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των διαφορετικών ε, δικτών αποτελεσμάτων, result indicators, και αν είναι δυνατόν με κάποιο τρόπο στο μέλλον να, βρεθεί, να καταλήξουν σε ένα ενιαίο σύνολο δικτών για όλε τις διαθέσιμε χρηματοδοτήσει. Διότι κάτι τέτοιο σίγουρα θα βοηθήσει. Τελευταία ερώτηση προ την Επιτροπή. Πώ προτίθεται να πιέσει τι χώρε μέλη να καταγράφουν τις προσπάθειές τους καταγραφής των αναγκών των πολιτών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή μια ε, προσέγγιση εκ των κάτω, διότι έχουμε εκπροσώπους των πολιτών που συχνά οι ανάγκες τους δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη, διότι οι συμφωνίες γίνονται μονάχα στο εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι χώρες μέλη κάνουν όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να εγγυηθούν την εκ των κάτω, bottom-up προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ Μαρτίνα. Μεγάλος αριθμός ερωτήσεων λοιπόν τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κοντά μας αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Πόπενς. Μπορείτε παρακαλώ να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μπάρκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το performance audit. Ευχαριστούμε το Ελεγκτικό Συνέδριο και διότι ανεγνώρισε σε ορισμένα σημεία το έργο της Επιτροπής. Είναι αληθές ότι ε, καθυστερεί ορισμένε φορέ η έγκριση προγραμμάτων και κάνουμε προσπάθειες να τα προλάβουμε και με ε, επιχειρηματικά προγράμματα και με συμφωνίες. Έχουμε αρχίσει και τον ανεπίσημο διάλογο με τις χώρε μέλη ήδη από την προηγούμενη περίοδο όταν κατανοήσαμε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά σε συνεργασία με τις χώρες μέλη επί της ουσίας των προγραμμάτων. Γιατί δεν γνωρίζαμε εξ αρχής ποια χρηματοδότηση θα πήγαινε σε ποια χώρα μέλο και για ποιο πρόγραμμα. Νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή απέδωσε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμα κάποια στοιχεία περιπλοκότητας, αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε την πολιτική συνοχή να δείχνει ότι η χρηματοδότησή μα, οι επενδύσει μα είναι στοχευμένε. Έχουμε αρχίσει και βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά απασχόληση και ανάπτυξη επιτόπου και στις περιφέρειες και στις χώρες μέλη. Το, η εκθέση του άρθρου 16 που ακούστηκαν εδώ για πρώτη φορά δείχνουν την επίτευξη των αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένου τομεί και προσπαθούμε ε, να συνοψίσουμε όλους αυτούς τους δείκτες ώστε να δείξουμε τι προσπαθούμε να επιτύχουμε με τα ταμεία μας. Αληθές είναι επίσης ότι έχουμε επενδύσει πολύ στην διαφάνεια και στο benchmarking και οι ανοιχτέ πλατφόρμες δεδομένων που υπάρχουν και που περιλαμβάνουν τι πληροφορίε και στο επίπεδο προγραμμάτων και στο επίπεδο προτεραιοτήτων, όπω είχε σχεδιαστεί όταν εγκρίναμε τα προγράμματα και τι οποίε επικαιροποιούμε διαρκώ τις πλατφόρμες Αυτέ επιτρέπουν κάποιο benchmarking ανάμεσα σε παρόμοια προγράμματα με παρόμοιε προτεραιότητε. Και ενθαρρύναμε τη μονάδα μα να χρησιμοποιεί τι πλατφόρμες δεδομένων και να, να υποβάλει στις ε, επιτροπές παρακολούθησης, monitoring committees. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι στην πράξη κάνουμε πολλά για να επιτρέψουμε την σύγκριση και το benchmarking. Νομίζω ότι τα βασικά σημεία κριτικής αναφέρονται ε, στις περιπλοκότητες. Θυμηθείτε όμως ότι η πολιτική μας είναι από μόνη της περιπλοκή. προωθούμε την συγκέντρωση για την Ευρώπη 2020 και παρόλα αυτά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη συγκεκριμένες εδαφικές αναγκαιότητες και προφανώς βγαίνει τελικώς το πλαίσιο των αποδόσεων πολύ περίπλοκο. Πάντως συνεργαζόμαστε διαρκώς με τις χώρες μέλη για να βελτιώσουμε το reporting μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο και με τα διάφορα ορόσημα και με τους διάφορους δείκτες που εντάσσονται στα προγράμματα. Επίσης είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε ετήσιες εκθέσεις απόδοσης και στέλνουμε σύνοψη και σε εσά και στο Συμβούλιο και σε όλους για το 2017 που είναι ένα ιδιαίτερο έτος διότι οι χώρες μέλη θα μας υποβάλουν εκθέσεις προόδου και στο τέλος θα υποβάλει η Επιτροπή ε, έκθεση στρατηγικής και ελπίζουμε ότι εκεί θα δείτε ορισμένες από τις ερωτήσεις σας να απαντώνται και θα δούμε επίσης και πώς αντιμετωπίζονται οι προτεραιότητες και πώς επιβάλλεται, πώς ενισχύεται η θεματική συγκέντρωση. Έχουμε αναζητήσει τις 10 προτεραιότητες και τις έχουμε προωθήσει που ανταποκρίνονται λίγο πολύ και στα όσα επενδύουμε στο προγραμμάτων μας αλλά έχουμε και κάνει και πολύ καλύτερη διασύνδεση και με το ρυθμιστικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό εξάμεινο και με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η μετανάστευση και ζητήματα επίσης ασφάλειας και άμυνας. Και είναι σημαντικό να θυμούμεθα ότι ο προγραμματισμός μας όπως είναι σχεδιασμένος μπορεί να είναι εύκαμπτος και μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τις νέες σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα μας τα προγράμματα. Το μόνο που θέλω να πω εκτός τούτων είναι ότι η performance, η βελτίωση της απόδοσης δηλαδή, ασφαλώς και αποτελεί προτεραιότητα για μας. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε επίσης για να συλλέξουμε τα αναγκαία δεδομένα και να κάνουμε τις αναγκαίες αναλύσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά το μέλλον, είναι σαφές νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει πρώτα να καταθέσει λευκή βίβλο για το μέλλον των χρηματοδοτήσεων, κάτι το οποίο θα είναι νομίζω διαθέσιμο, δηλαδή το Λευκό Βιβλίο ήδη από τούτη εδώ την εβδομάδα και θα αποτελέσει την βάση συζητήσεων για πολύ συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτά θα ήθελα να πω για την ώρα, αλλά θα επανέλθουμε βεβαίως ε, επί το συγκεκριμένο περιεχομένο της εκθέσεως στα τέλη του έτους και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι όντως έχουμε μια προσέγγιση hands-on για την εφαρμογή των προγραμμάτων μας. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν πετύχαμε απλούστευση. Για το ERDF έχουμε μείωση 50% του αριθμού των προγραμμάτων. Έχουμε και πολλές χώρες μέλη που, όπως οι βαλτικές χώρες αλλά και άλλες που εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα, έχουμε και άλλες χώρες όπου η διοργάνωσή τους είναι πολύ περίπλοκη, όπως η Αυστρία. Αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να συμβόμαστε και το γεγονός ότι ορισμένες χώρες μέλη κάνουν και πολύ σημαντικές περιφερειακές μεταρρυθμίσεις δίνοντας μεγαλύτερες εξουσίες στις περιφέρειες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία και η Ελλάδα. Και αυτό οφείλουμε να το λάβουμε σοβαρό, υπόψη όταν καταστρώνουμε τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Εν το συνόλο νομίζω ότι έχουμε πετύχει μια καλή αρχιτεκτονική διαμόρφωση των προγραμμάτων μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε και για το μέλλον, αλλά δεν υπάρχει και καμία λύση που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί κάθε χώρα μέλος είναι και διαφορετική. Ευχαριστώ. Οι περισσότερες ερωτήσεις απευθύνονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τόσο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά αν θέλετε μπορείτε να κάνετε κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. No, I explain our observation in my opening speech. But uh, like to add that uh, uh, Ήδη ανέφερα κάποια πράγματα κατά την ε, ανακτήρια μου παρέμβαση, αλλά, αλλά όπως ε, ε, θα διαπιστώσατε η δική μου έκθεση είναι πιο θεωρητική αν θέλετε και όχι τόσο πρακτική. Πρόκειται δηλαδή μία βάση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των ταπανών των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, η δική μου τοποθέτηση αφορά το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα στο μέλλον και ειδικότερα ποιος θα είναι αντίκτυπος του Brexit. Γιατί όλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι αφορά δηλαδή τον προπολογισμό, θα μεταβληθούν και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ε, μία δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω και στο οποίο ήδη αναφέρθηκα είναι ότι βρισκόμαστε στα τελικά στάδια διατύπωσης των ε, υπαριθμών δύο, ας πούμε, νέα έκδοση, αν θέλετε, των συμφωνιών εταιρική ε, σχέση. Και εκεί θα ασχοληθούμε ακριβώς με τα ζητήματα εκείνα που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά στο πλαίσιο αυτών των ε, συμφωνητήων εταιρικέ σχέσει, δηλαδή ειδικότερα το αποθεματικό τη ε, απόδοση και ε, της, των προτέρων αιρεσιμότητε. Νομίζω πω αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα γίνει με την Επιτροπή και όπως σας είπα εδώ, ο στόχος της έκθεσης είναι να δημιουργήσουμε και μία βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωθεί η μελλοντική δαπάνη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν από την πλευρά μου σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Πρινίστη, θέλετε πάλι το λόγο για να κάνετε κάποια τελικά σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, τελικά σχόλια προς το παρόν, γιατί θα πούμε ακόμα πολλά για αυτό το θέμα. Πάντως, ε, θεωρώ πως οι απαντήσεις του αναπληρωτή διευθυντή είναι ενδιαφέρουσες και να πω τα εξή. Να δούμε καταρχήν τα θετικά στοιχεία. Δηλαδή η πρακτική που ακολουθείται σε ό,τι αφορά τις άτυπες διαπραγματεύσεις ε, πριν από την έναρξη της τρέχουσας ε, περίοδου. Ναι. Ε, νομίζω πως αυτό ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις που έκανε η Μαρτίνα Λαβαγιώβα και τα όσα είχαν αναφερθεί ήδη στο παρελθόν. Σε σχέση με αυτό το σημείο, εγώ λοιπόν θα παρότεινα την Επιτροπή όχι μόνο να επαναπαυθεί στα όσα έχει επιτύχει μέχρι τώρα, αλλά ενδεχομένως να ξεκινήσει να ε, εκπονεί ένα σχέδιο κρίσης, αντιμετώπισης κρίσης, γιατί θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την προετοιμασία ε, του νέου ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου να γίνουν πολλά πράγματα την τελευταία στιγμή, ε, διαπραγματεύσει την τελευταία στιγμή, τη τελευταία ώρας και ούτω καθεξής. Οπότε, νομίζω πως αυτή η πτυχή ε, παραγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την Επιτροπή. Ε, όταν μας λέει απλώς και, εμένα, απλώς και μόνο ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι θα έρθουμε με τις προτάσεις μας, μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση γιατί κατά πάσα πιθανότητα τελικά η κατάσταση την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και ένα πόρισμα το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ είναι ένα που, το οποίο αναφέρεται και στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου αλλά και αναφέρεται από την Επιτροπή. Ότι δηλαδή οι αυξημένες αρμοδιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά κάποιον τρόπο αποτελούν τροχοπέδι γιατί για παράδειγμα δημιουργούν περισσότερες καθυστερήσεις. Όχι. Δηλαδή ποια είναι η λύση ε, για αυτό το πρόβλημα. Να μειώσουμε τις αρμοδιότητε τις εξουσίες του Κοινοβουλίου σε αυτό το τομέα. Αυτή είναι η λύση. Ε, πρόκειται δηλαδή για μια τρομακτική παρανόηση. Και σίγουρα θα πρέπει να διασφαλιστούν αυτές οι εξουσίες που έχει το Κοινοβούλιο και από εκεί και μετά να γίνουν προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη εκτέλεση σε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν και πάλι εδώ το χρονοδιάγραμμα, έχουμε κάποιε ενθαρρυντικέ ενδείξει από την πλευρά τη Επιτροπή, αλλά παραμένουν μία σειρά από ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την απλούστευση, και στο οποίο αναφέρθηκε και η Ματίνα, ο αναπληρωτή ε, διευθυντή μα είπε ότι το αρνείται ουσιαστικά. Ότι δηλαδή όχι, επιτύχαμε απλούστευση από την πλευρά τη Επιτροπή. Αλλά αυτό είναι περίεργο γιατί ο τίτλος της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου τι λέει. Και στο συγγνώμη που θα σας ε, σπαταλήσω ένα-δύο χρόνια από το σχόλιο σας, ε, Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά το πρόγραμμα εμφανίζει έναν υψηλότερο δείκτη περιπλοκότητας. Οπότε η Επιτροπή λαμβάνει στα σοβαρά υπόψη της αυτή την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου ή όχι. Και ένα τρίτο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξή. Εφιστώ την προσοχή σας και εκφράζω την ανησυχία μου ω προ το εξή. Ανέφερε λοιπόν αυτού τη διευθυντή τη νέα προκλήση ό,τι αφορά τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την άμυνα και ούτω καθεξή. Η πολιτική όμως συνοχή δεν αφορά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η πολιτική συνοχή είναι μια μακροπρόθεσμη ε, στρατηγική, σε βάθος χρόνου, αν θέλετε, που θα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα έργα. Και βέβαια για την υλοποίηση αυτών των στόχων χρειαζόμαστε και ένα πολύ καλά διατυπωμένο σχέδιο. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει και ένα αντίστοιχο ψήφισμα από τη δική μας πλευρά. Πρόεδρος, ε, ναι, ευχαριστούμε τον κύριο Πυρίνσκι. Θα ήθελα και εγώ να κάποια να κάνω και εγώ κάποια σχόλια, γιατί συμμετέχω όχι μόνο σε αυτή την Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή που ασχολείται με την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ε, και να πω ότι ε, γνωρίζουμε ως κράτη-μέλη ότι όλοι αξιοποιούμε τα κονδύλια ε, εδώ από την πολιτική συνοχή και γνωρίζουμε πως σε δημοσιονομικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο πρόκειται ακριβώς για τα πιο σημαντικά ε, τα ταμεία για τα πιο σημαντικά κανδύλια. Και ε, αυτά τα project, δηλαδή τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, είναι εκείνα που γνωρίζουν στο μεγαλύτερο βαθμό οι πολίτε μα. Οπότε κάθε είδου επικοδομητική κριτική την οποία ασκούμε, ε, την ασκούμε ακριβώ επειδή θέλουμε να βελτιωθεί και στο μέλλον αυτή η πολιτική συνοχή. Θέλουμε δηλαδή να παίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του, των πολιτών δημοσιονομικών πλαισίων. Θέλουμε να εκτελείται στο ταχύτερο δυνατό από την πλευρά τη Επιτροπή. Θέλουμε να είναι η πολιτική αυτή όσο το δυνατόν τον απλούστερη. Θέλουμε να ε, είναι πιο στοχευμένη σε ό,τι αφορά δηλαδή την, ε, τις επιδόσεις και, τις, ε, και τους συγκεκριμένους στόχους. Και από εκεί και μετά γνωρίζουμε βέβαια πως υπάρχουν εκείνοι που είναι επιφυλακτικοί, που αμφισβητούν, που θεωρούν για παράδειγμα ότι ενδεχομένως δεν χρειάζεται να επενδύονται τόσα κονδύλια ε, και ούτω καθεξής. Οπότε εμεί θα πρέπει να καταδείξουμε σε αυτούς που αμφισβητούν την πολιτική συνοχή ότι έχει πολλά να προσφέρει και στο μέλλον να ε, ε, δώσει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα προ όφελο των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ο στόχο μου, ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την πολιτική συνοχή και στο μέλλον. Οπότε όποια σχόλια κάνουμε, σα παρακαλούμε να τα εκλάβετε ε, με αυτόν τον τρόπο από την πλευρά μα. Α κλείσουμε λοιπόν με αυτό το σημείο και α περάσουμε στο σημείο 4 τη σημερινή διάταξη και πάλι εδώ αρμόδιο συζητητή ο κύριο ε, Γεωργή Πυρίνσκι, αλλά προτού του δώσω το λόγο για να αναφερθεί στην ειδική έκθεση, να ότι πρόκειται για ε, την προστασία του προπολογισμού από τι παράτυπε δαπάνε και πρώτα θα δώσω το λόγο λοιπόν στον αρμόδιο εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Κρέτα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγητά, βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη μου ευχαρίστηση να σα παρουσιάσω την ειδική μα έκθεση 4 του 2017 για την προστασία του προπολογισμού τη Ένωση όσον αφορά τι παράτυπε δαπάνε, όσον αφορά την πολιτική τη συνοχή. Ο ε, βασικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εξασφαλίσει ότι ο προπολογισμό εκτελείται σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί και προβλέπονται σε κανονισμού και διατάξει γενικότερα. Οπότε έχουμε εδώ πέρα δύο μέσα. Τα μέσα, τα πρόληπτικά, ούτω ώστε να μην υπάρχουν παράτυπες ε, δαπάνες πριν γίνουν δηλαδή εκταμιεύσεις και επίσης έχουμε και τις δημισιονομικές διορθώσεις προστατεύουν τον ε, προϋπολογισμό από το βάρος των λανθασμένων ταπανών και έτσι αποκαθίσατε μια κατάσταση ε, ούτω ώστε να είναι τα πράγματα όλα σύντορα και ε, να συμμορφώνονται προς τους κανόνες. Κατά τον οικονομικό έλεγχο αξιολογήσαμε το κατά πόσον αυτά τα δύο μέσα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούσαν κάποιες συγχρηματοδοτήσεις και κάποιες παράτυπε δαπάνε στην ε, πολιτική της συνοχής. Μιλούμε για 350 δις ευρώ για τις ε, χρήσεις 2017 έως 2013 και 2014-2020. Μιλούμε δηλαδή για το 1 τρίτον του συνόλου του προηγουμένου της Ένωσης και συνολικά διαπιστώσαμε ότι αποτελεσματική χρήση των μέτρων ε, ίσχυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2007 με 2013 <clears throat> για να προστατεύσει τον προηγούμενο της Ένωσης από παράτυπες δαπάνες. Ε, είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποια προληπτικά μέτρα, αλλά ε, και δημοσιονομικές διορθώσεις περισσότερο στην περίοδο 2013 περισσότερο παρά την προηγουμένη περίοδο και έλαβε κάποια μέτρα τα οποία αναλογικό χαρακτήρα και είχε στόχο και επικεντρώθηκε στα πιο ρηψοκίνητα κρατημέλη. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίεσε τα κρατημέλη να αντιμετωπίσουν τι αδυναμίε διαχείριση, τα στήματα ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, πάνω κάποια προβλήματα που ε, είναι το ότι δηλαδή τα μέτρα αυτά είναι τόσο περίπλοκα ότι χρειάζεται χρόνο τόσο ώστε κανεί να μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό ρίσκο για τα κράτη-μέλη, Οπότε το πρώτο θέμα είναι το κατά πόσο τα πράγματα γίνονται σωστά από τα κράτη-μέλη και αν ε, δεν υπάρχει κάποιο είδου παράτυπη δαπάνη, τότε μπορεί να κάνει και τα προληπτικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, διαπιστώσαμε ότι είχε δυσκολίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο τη υλοποίηση των δημοσιονομικών διορθώσεων, ε, γιατί πολλέ φορέ η ενημέρωση και οι πληροφορίε από τα κράτη-μέλη δεν βοηθούσαν. Τώρα όσον αφορά τι εκθέσει Ευρωπαϊκή για τα προληπτικά μέτρα και τι δημιουργικέ διορθώσει, διαπιστώσαμε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει μια γενικότερη εποπτεία τη κατάσταση, διότι τα στοιχεία και οι πληροφορίε ε, κατανέμονται σε περισσότερα έγγραφα και δεν υπάρχει κάποιο είδου συγκέντρωση αυτών των στοιχείων. Επίση, θεωρήσαμε ότι εμπλεκόμενο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα θυμάστε ότι είχατε περάσει και εσείς από κάποιες ε, συνεντεύξεις και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους οι εκθέσεις Επιτροπής δεν περιέχουν αρκετά στοιχεία όσον αφορά συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών και καλών πρακτικών σε σχέση με το πώς γίνεται η πρόληψη, η ανείχνευση και η διόρθωση των επαναλαμβανομένων προβλημάτων. Οπότε θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ποιο είναι το σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ως αρμοδιότητα να ελέγχει και να ε, διατυπώνει κάποιε συστάσει, αλλά δεν μπορεί να συμβουλεύσει άμεσα τα κρατημένη. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αντίθεση με εμά, κάνει οικονομικού ελέγχου συχνότερα. Άρα είναι στέση περισσότερο από εμά να μπορέσει να διαπιστώσει κάποιε ε, να προδεί μάλλον σε κάποιε συστάσει για τη βελτίωση τη λειτουργία του συστήματο του δημιουργικού ελέγχου και της διαχείρισης. Τώρα, όσον αφορά τι κανονιστικέ νομοθετικέ διατάξει του 2014-2020 διαπιστώσαμε ότι υπάρχει βελτίωση όσον αφορά το σχεδιασμό του συστήματο και έτσι έχει τώρα περισσότερε αρμοδιέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί τώρα να δει το ότι δεν έχουμε παράτυπε δαπάνε από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και έτσι τώρα μπορεί καλύτερα να προστατεύσει αυτόν τον προπολογισμό η Επιτροπή. Τέλο, θέλω να επισύρω την προσοχή σα στο ότι έχουμε διατυπώσει κάποιε συστάσει αυτή μα την ειδική έκθεση και συνιστούμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέχει να μην γίνονται λάθη όσον αφορά τι εκταμιεύσεις και τι πληρωμέ. και θα πρέπει επίση να βελτιώσει του ελέγχου και τι διαδικασίε με την υποβολή εκθέσεων και έτσι να χρησιμοποιήσει τις νεες αρμοδιοτητε αρμοδιότητες περίοδου 14-20 και σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εμείς για τα όσα μας είπατε. Και τώρα στον εισηγητή τον κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Και πρώτα πρόκειται σαφώς για επιτυχημένη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής που αρχίζει με έγκαιρο προγραμματισμό αλλά μπορεί να αποδειχτεί επιτυχής όπως είπατε και πριν μόνο εφόσον σέβεται τις αρχές της υγιούς δημοσιονομικής στρατηγικής. Και αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπαριθμών 4 προβλέπει μέτρα και διορθώσεις και για περαιτέρω βελτιώσεις του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών μελών για την προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης εκφράζω τη βαθιά εκτίμησή μου και τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Γκρέτεν και στην ομάδα του για την πραγματικά θαυμάσια δουλειά που έχουν κάνει με την ειδική έκθεση. Και θα ήθελα ε, να καλωσορίσω και την αποδοχή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου και αναμένω να τα εφαρμόσει πλήρω και στον δέοντα χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της για να προστατεύσει τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Έχει, κάνει, έχει λάβει και διορθωτικά μέτρα και μάλιστα πολύ νωρίτερα από ότι στην περίοδο του 2000-2006 και με μεγαλύτερα αποτελέσματα. Θετική τάση λοιπόν που θα πρέπει να συνεχιστεί και στην υπόλοιπη προγραμματική περίοδο και προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει τις συστάσεις του ελληνικού Συνεδρίου προκειμένου και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να αγρυπνήσει ό,τι αφορά την εφαρμογή του προπολογισμού και στο μέλλον. Θα πρέπει επίση να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει αναλυτική έκθεση για όλα τα προληπτικά μέτρα και διορθώσεις που έχει κάνει για την περίοδο 2007 έως 2013 στην βάση της εκθέσεως που έχει υποβληθεί για την προηγούμενη περίοδο το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τι διορθωτικές ε, διορθώσεις θα πρέπει να ενισχυθεί, λέει και το ελληνικό συνέδριο. Ο βασικός στόχος θα πρέπει όμω να παραμείνει η πρόληψη των παρατυπιών. Και θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δυνατόν συντομότερο να φτιάξει ένα σύστημα παρακολουθήσης το οποίο θα επιτρέπει ε, συγκριτικές αναλύσεις και για προληπτικά μέτρα και για διορθώσεις για την περίοδο 2014 έως 2020. Τα άλλα θεσμικά όργανα και οι αρχές των χωρών μελών θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στις προφορίες αυτές. Έχουμε κάποια πρόσθετα σχόλια και συστάσεις στο έγγραφο εργασίας, καθώς και συμμεράσματα και παρατηρήσεις και όπως σωστά λέει το ελεγκτικό συνέδριο, διακοπές χρηματοδοτήσεων και αναστολές αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τις χώρες μέλη. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ισορροπημένες προσπάθειες για την προστασία του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής της συνοχής, αναγνωρίζοντας την ανάγκη έγκυρης εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Είναι σημαντικό επίσης οι χώρες μέλη να εντοπίζουν παρατυπίες και να κάνουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και να δίνουν και χρόνο, περισσότερο χρόνο για την επίλυση των προβλημάτων. Επομένω και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη ε, να είναι πιο ενεργές, πιο δραστήριες και υπεύθυνε ε, να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν τις παρατυπίες, να εφαρμόζουν ελεγκτικούς μηχανισμούς στις επικράτειές τους και επιπροσθέτω πρέπει να ζητήσουμε από τι χώρε μέλη να χορηγούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκή και σε ποσότητα και σε ποιότητα ε, ευρωπαϊκής όγκους πληροφοριών για να μπορούν να ικανοποιούνται και οι διαδικασίε χωρίς έξτρα γραφειοκρατική επιβάρυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως θα πρέπει να τους προσφέρει ρυθμιστική ασφάλεια και συνεργασία και βοήθεια για να τους επιτρέπει να διατυπώνουν τις ανάγκες τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές των χωρών μελών για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων πρώτου και δεύτερου επίπεδου και θα πρέπει να δίνει και κατευθύνσει στις χώρες μέλη για τις οριζόντιες εκθέσεις που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διορθώσεων που θα έχουν κάνει οι χώρες μέλη, που κάνουν οι χώρες μέλη οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου θα επιτρέψουν στο μέλλον να εντοπιστούν οι συστημικές αδυναμίες και να βελτιωθεί η λειτουργία του συνολικού συστήματος. Τέλος, δύο ερωτήσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή, ως εξής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνέδριο βρήκε ενδείξεις για τις διορθώσεις και για το 2007-2013, για την περίοδο 2007-2013. Ομιλώ για την παράγραφο 11. Αν μπορεί να επεκταθεί λίγο σε αυτό, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Έως τώρα δεν έχουν ληφθεί αποφάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οικονομικές διορθώσεις για το 2007 έως 2013, την προγραμματική περίοδο των ετών αυτών. Και μιλώ για την παράγραφο 57. Μήπως μπορούν να επεκταθούν λίγο και εκεί. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι. Ισκιώδης. Αντρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω τον ε, φίλο Πυρίνσκι για την αποσίωση και σκληρή δουλειά και για την έγκαιρη έκθεση. Τώρα μάλιστα που γίνεται και το φόρουμ για τη συνοχή. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή είναι μια μακροπρόθεσμη πολιτική επενδύσεων και χρειάζεται προστασία του προπολισμού. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα. Όμως, η μείωση των οικονομικών διορθώσεων δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μειωθεί η αναγκαιότητα για δημοσιονομικές διορθώσεις, ώστε να μην προκαλέσουμε έξτρα επιβάρυνση και στο τοπικό, περιφερειακό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορα βήματα. Ένα από αυτά είναι να βάλουμε πιο συγκεκριμένους δείκτες και στόχους στην εκ των προτέρων ανάλυση των, των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη εικόνα, πιο καθαρή εικόνα για τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Από την άλλη μεριά περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα στις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης επιτρέπουν καλύτερη κατανόηση των αναγκών των τοπικών φορέων. Εάν βάλουμε δηλαδή ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχων και λογοδοσίας, θα διευκολύνουμε και τη ζωή των δικαιούχων. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι περισσότερες παρατυπίες οφείλονται σε σφάλματα, όχι σε πρόθεση απάτης. Άρα χρειάζεται περισσότερη τεχνική υποστήριξη που ίσως να ε, μειώσει την αναγκαιότητα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων. Τέλος, θέλω να συγχαρώ την ομάδα BCA για την έκθεση, παρόλο που η περίοδος στην οποία αναφερόμαστε είναι εδώ και μια δεκαετία, έχουμε εκθέσει συνοχής ανά Έτσι ε, θα πρέπει να συνεχίζουμε με τις του ελεγκτικού συνεδρίου. Γιατί αυτό θα μας επιτρέψει και επιτάχυνση της ε, αν αποφασίσουμε, αν, αν γνωρίζουμε προς τα που κινούνται τα επιχειρησιακά προγράμματα. και αν μπορούμε να κάνουμε και εγκαιρότερα την ανάλυση αυτή, αλλά όχι 2008-2009. Η Μαρτίνα, ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστώ το Ελληνικό Συνέδριο για το καλό συνταγμένο έγγραφο με τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Για μας, τους προστάτες του προϋπολογισμού, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έγγραφο εργασίας. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Αντρέη, διότι αναγνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ορθή χρήση των εργαλείων που διαθέτει για την περίοδο 2007-2013. Αλλά εάν οι χώρες μέλη εντοπίζουν παρατυπίες και λαμβάνουν έγκαιρα προληπτικά μέτρα, θα χρειάζονται λιγότερες διορθώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό νομίζω ότι θα καταστήσει την διαδικασία και πιο αποτελεσματική αλλά και πιο οικονομική. Άρα όχι μόνο οι χώρες μέλη, αλλά και, όχι μόνο και οι Κομισιόν, και οι χώρες μέλη πρέπει να λαμβάνουν προληπτικές ενέργειες όχι μόνο για το cash flow, αλλά και σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους και την έγκαιρη απόλυψη των χρημάτων. Άρα πρέπει οι χώρες μέλη να φανούν πιο υπεύθυνες. Θα ζητήσω από το Ελληνικό Συνέδριο και την Κομισιόν να δώσουν κάθε δυνατή υποστήριξη και κατευθύνση στις χώρες μέλη. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην προηγούμενη έκθεση, ότι θα πρέπει να διδαχτούμε από τα παλαιότερα σφάλματά μας και θα πρέπει να μειώσουμε τα προσδιόρθωση ποσά. Ας αντλήσουμε επιτέλους τα αναγκαία διδάγματα. Μου άρεσε επίση η σύσταση του Ελληνικού Συνεδρίου που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τα συστήματα παρακολούθηση, τα οποία πράγματι πρέπει να ολοκληρωθούν. Να περιλάβουν και την financial correction με καλύτερε συγκριτικέ αναλύσει. Έχω και μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν είμαι βέβαια εάν το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να απαντήσει. Διότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην παράγραφο 8, εκεί περιλαμβάνεται ένα ποσοστό απορρόφηση στο τέλος της προγραμματικής περίοδου τη τάξη του 65%. Όπου φτάνει όμως σε λιγότερο από το μισό, ενώ ήταν 20% στο 2010. Και το ίδιο σενάριο απορρόφησης εμφανίζεται σε όλες τις προγραμματικές περιόδους. Ποια είναι η άποψη του Ελληνικού συνεδρίου. Όσο πιο πολύ παρατείνεται η απορρόφηση, τόσο περισσότερο σε σφάλματα υποπίπτει ε, ε επένδυση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε τώρα, μπορούμε να το συζητήσουμε και άλλη φορά. Είδα αυτό το νούμερο και μου κίνησε το ενδιαφέρον έχει και κάποια σχέση εδώ με μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βελτίωση της απορροφητικότητας όταν προγραμματίζει την προγραμματική περίοδο. Μιλώ πάντα για αυτό το ποσοστό απορρόφησης. Thank Σας ευχαριστώ. Έγιναν κάποια ερωτήματα λοιπόν στην ε, Επιτροπή. Οπότε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζίμπερτ από την Επιτροπή ο οποίο είναι ο Διευθυντής Ελέγχων τη Γενική Διεύθυνση ε, Ρέτζιο. Ο λόγος σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέδεν και την ομάδα του για αυτήν την ε, διεξοδική έκθεση. Και ευχαριστώ και τον κύριο Πυρίνσκι για ε, τα συμπληρωματικά σχόλια που έκανε σε σχέση με την έκθεση, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτές τις συστάσεις και χαιρετίζουμε και εμείς το γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση του συνεδρίου επιβεβαιώνει τα όσα εμείς έχουμε αναφέρει κατά την ε, διάρκεια των τελευταίων ετών εδώ στην Επιτροπή σας ότι δηλαδή έχουμε βελτιώσει την χρήση των νομικών εργαλείων ως Επιτροπή σε ό,τι αφορά ε, και τις ε, διορθωτικές και τις αποτρεπτικές, οι προληπτικές αν θέλετε πτυχές. Ε, θυμάμαι δηλαδή τα όσα είχαμε συζητήσει την περίοδο 2008-2009 εδώ σε αυτή την Επιτροπή και διαπιστώνουμε πόσο έχουμε προχωρήσει έκτοτε και ε, όπως ανέφερε και το ελεκτικό συνέδριο έχουμε ήδη βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά ε, σφαλμάτων σε σύγκριση με το 2006 και ήδη έχουμε σχετικές ενδείξεις για το 2013. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι ε, το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει για το 2020 με περισσότερες ε, ευθύνες, με την ευθύνη δηλαδή των κρατών μελών στην καρδιά του, θα ανταποκριθεί στα αυτά που αξιώνεται, δηλαδή ε, στην ανάγκη του να ε, αποτρέψουμε αν θέλετε την εμφάνιση λαθών ε, από την αρχή, όχι δηλαδή την αντιμετώπιση εφόσον έχουμε εμφανιστεί. Γι' αυτό λοιπόν το νέο μας σύστημα σε σχέση με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές έχουμε αλυσίδες, το σύνολο της αλυσίδας ελέγχων ε, το, η οποία θα πρέπει να ε, ολοκληρώνεται στα κράτη-μέλη και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον υπολοιπόμενο κίνδυνο ε, όπως αυτός θα επαληθεύεται στο τέλος κάθε σε σχέση με τους ονοκολογαριασμούς. έχουμε ήδη δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση σε ό,τι αφορά τις αιτήσιες δράσεις και πραγματικά διαπιστώνουμε ότι το νέο σύστημα μας επιτρέπει, επιτρέπει να διαπιστώνουμε ποιο είναι το υπόλοιπο, αν θέλετε, των σφαλμάτων που υπάρχει, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε ποιε είναι τελικά οι διορθώσεις που είναι απαραίτητες για κάθε χρόνο. Πάντως, συμφωνώ απολύτως μαζί σας αυτό που είπατε, ότι ο στόχος δεν είναι να αξιοποιεί τέτοιου είδους εργαλεία επιτροπή, ο στόχος είναι τα κράτη-μέλη να ασκούν μια όσο το δυνατόν πιο προληπτική ε, ε, πολιτική σε ό,τι αφορά τα, τα σφάλματα αυτά. Ε, και εδώ να σας παραπέμψω και μια σχετική έκθεση που έχουμε σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις και όπου έχουμε αναφέρει ένα αθρηστικό επίπεδο διορθωτικών ε, διορθώσεων ύψους 2,9 δις ευρώ με βάση τα δικά μας προγράμματα και από εκεί και μετά τα ίδια τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε ε, ως διορθώσεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια διορθώσεων για τα κράτη-μέλη και όπως ε, ε, είπατε και εσείς εδώ ο στόχο είναι να υπάρξει καλύτερη πρόληψη λανθών, λανθών σφαλμάτων από πλευρά των κρατών μελών. Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε πράγματι εκπονήσει καθοδήγηση από δική μα πλευρά και μάλιστα αναφέρθηκε ήδη και από την ε, κυρία ε, Λαμπάνοβα, ότι έχουμε δηλαδή εκπονήσει ενδεχομένω ε, υπερβολικέ ε, οδηγίε, υπερβολικό αριθμό οδηγιών με 2.500 σελίδε και όπου περιλαμβάνονται οδηγίε σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη δειγματοληψία από την πλευρά των διαχειριστικών αρχών και ούτω καθεξή. Όμως ο στόχο είναι ακριβώ εδώ να παράσχουμε βοήθεια στις αρμόδιες αρχέ των κρατών μελών προκειμένου να αποφεύγουν την, ε, τα ασφάλματα. Και έχουμε παρουσιάσει εδώ στην ε, ε, Επιτροπή, βασιζόμενη ακριβώς και αυτές τις εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, στοιχεία σε ό,τι αφορά ακριβώ ε, τα σφάλματα που γίνονται και στον τομέα, για παράδειγμα, των δημοσίων συμβάσεων. Εδώ δηλαδή προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα πιο κοινά ε, σφάλματα, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να τα αποφεύγουν και επίσης έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων, peer-to-peer, ε, για να μπορούν να βοηθούνται τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Γιατί ένα πράγμα είναι η Επιτροπή ε, άνωθεν, θέλετε, να ε, αναφέρει στα κράτη-μέλη το τι κάνουν λάθος και άλλο είναι τα ίδια τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους και να βλέπουν ποια είναι τα προβλήματα. Από εκεί και μετά ε, συμφωνούμε πλήρως με τις ε, τέσσερις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση και ε, σας διαβεβαιώ ότι σε αυτή τη φάση εξετάζουμε τις δηλώσεις κλεισίματος στο πρόγραμμα των περίοδος του 2013 και έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή να μην κλείνει προτού διασφαλίσει ότι έχει φτάσει στο επίπεδο σφάλματος μπυλό όπως λέγεται. Και ε, σε αυτό ακριβώ το πλαίσιο ζητούμε συμπληρωματικού ελέγχου από τα κρατημέλη, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να κλείνουμε τα προγράμματα με ε, ένα μη ουσιαστικό, δηλαδή με ένα επουσιώδες αν θέλετε επίπεδο σφαλμάτων. Τώρα σε ό,τι αφορά τις εστάσεις για τα κρατημέλη, ναι, συμφωνούμε ότι δηλαδή η υποβολή εκθέσεων τελικά είναι κατακαιρματισμένη, δηλαδή τα, τα, οι αναφορές είναι κατακαιρματισμένες σε διαφορετικές εκθέσεις. Έχουμε ε, την έκθεση ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προστασία των οικονομικών ε, ε, συμφερόντων της Ένωσης και πλέον αυτή για παράδειγμα η έκθεση έχει τώρα συγχωνευτεί σε μια ετήσια έκθεση MPR όπως λέγεται έτσι ώστε ακριβώς τα στοιχεία της, των επιδόσεων και τα στοιχεία της συμμόρφωσης να περιλαμβάνονται σε κοινή έκθεση σε ό,τι ακριβώς αφορά τις προληπτικές και διορθωτικές δράσεις της Επιτροπής. Τώρα σε ό,τι αφορά την παράκληση να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση και ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης από την πλευρά της Επιτροπής. Αναγνωρίζουμε σε κάθε ε, περίπτωση ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το υφιστάμενο ε, σύστημά μας ε, και αυτό γιατί στην αρχή είχαμε αναπτύξει διαφορετικά συστήματα για διαφορετικούς σκοπούς. Και εδώ έγινε και μία πολύ ε, χρήσιμη σύσταση της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου σε ό,τι αφορά την απλούστευση σε ζητήματα ελέγχου ε, και η οποία ακριβώ ανέφερε, αναφερόταν στην ανάγκη καλύτερων αναλύσεων και αναλύσεων οι οποίες θα αφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε όλοι να μπορούν να μαθαίνουν από τα λάθη που γίνονται χωρίς να χρειάζεται να κατονομάζουμε το ένα ή το άλλο κράτο μέλος πρόγραμμα. Όμω, είναι πολύ αποθαρρυντικό το να διαπιστώνουμε ε, ε, όταν βλέπουμε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, και εδώ αναφέρομαι και στη δική σας χώρα κύριε Πυρίνσκι, όπου έχουμε διεξάγει επιχειρησιακό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τον άξο 1 ε, και μετά έχουμε για παράδειγμα, ε, τον επόμενο χρόνο προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τον ίδιο άξονα, αλλά τελικά στο δεύτερο χρόνο όλα τα προβλήματα που είχαμε στον πρώτο άξονα προτεραιότητα επαναλαμβάνονται στο δεύτερο χρόνο. Οπότε ε, βλέπουμε ότι οι εμπειρίε, τα όσα δηλαδή μαθαίνουμε, τα διδάγματα δεν ε, γίνονται γνωστά σε όλου. Οπότε αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο μα να υπάρχει δηλαδή γνωστοποίηση αυτών των διδαγμάτων σε όλου, Δηλαδή να μην μαθαίνουν όλοι βέλτιστες μόνο πρακτικέ, αλλά να ακούνε και ποια είναι τα προβλήματα, ποιε είναι οι κακές πρακτικές του παρελθόντος, ποια είναι τα σφάλματα του, ώστε όλοι να μπορούν να μάθουν από αυτά. Και εγώ θα συζητήσω αυτό το ε, ζήτημα και με του εκπροσώπου των κρατών μελών στη συνάντηση που θα έχουμε στα μέσα Ιουλίου, ώστε να δούμε ακριβώ ποιο θα είναι ο καλύτερο τρόπο για να ε, διαδοθούν καλύτερα αυτές οι πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών. Τέλος, σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο σε ό,τι αφορά τις ε, ε, καθαρές διορθώσεις, καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις και εδώ έχουμε διαπιστώσει ότι για το 2013 τέτοιου είδους δημοσιονομικές διορθώσεις αν έχουν γίνει από την πλευρά των κρατών μελών μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και γι' αυτό θα είδατε και στην έκθεση ότι δεν λήφθηκε και μια σχετική απόφαση γιατί έως το 2013 Ε, είχαν τη δυνατότητα να προβαίνουν ε, από τις πλευρά στις δημοσιονομικέ διορθώσεις ε, Και εφόσον δηλαδή ήταν σε θέση να επιλύσουν τα σχετικά προβλήματα, είχαν τη δυνατότητα τα εν λόγω κονδύλια τους φάντους να τα αξιοποιήσουν. Τώρα, στον ε, νέο διομοσιονομικό κανονισμό προβλέπεται ότι ακόμα και αν το κράτος μέλος συμφωνήσει ε, στη διόρθωση, αλλά διαπιστωθεί αυτό ε, πολύ αργά, δηλαδή έχουν υποβληθεί όλες οι σχετικές εκθέσεις και έχουν κλείσει οι σχετικοί απολογισμοί, και διαπιστώνεται από την Επιτροπή σημαντικό πρόβλημα, μια σημαντική έλλειψη όπως προβλέπεται στον κανονισμό και από τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός. Ακόμα λοιπόν και αν το κράτος μέλο, ε, συμφωνήσει με τι διορθώσει που προτείνει η Επιτροπή, θα είναι υποχρεωμένο το κράτο μέλο να προβεί σε μια καθαρή διόρθωση ε, δημοσιονομική, net financial correction. Νομίζουμε πω αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ένα περαιτέρω ένασμα στα κράτη-μέλη να ολοκληρώνουν σωστά ε, το κρίσιμο των λογαριασμών σε αιτήσια βάση. Από εκεί και μετά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε ήδη ότι κάποια κράτη-μέλη δεν τολμούν να δηλώσουν τις δαπάνες τους γιατί φοβούνται ακριβώς το ενδεχόμενο του να προκύψει αυτή η καθαρή δημοσιονομική ε, διόρθωση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τελικά να δαπανούν πολύ χρόνο ε, σε ό,τι αφορά την τελική υποβολή των, ε, δεδομένων τους. Πράγμα βέβαια το οποίο έχει κακές επιπτώσεις, αντικές επιπτώσεις στην, στο ρυθμό εκτέλεσης των προγραμμάτων. Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι και μια αντική συνέπεια. Τέλος, θα ήθελα να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν ε, ε, περισσότερα διδάγματα από την περίοδο του 2013. Δηλαδή να, να μοιραστούμε τα διδάγματα, τα, τα, μεταξύ των κρατών μελών ε, και όταν θα έχουμε ολοκληρώσει πλήρω το κλείσιμο του 2013, ακριβώ αυτό θα κάνουμε. Είμαστε δηλαδή σε κάθε περίπτωση διατεθειμένοι να απευθυνθούμε στου ε, συναρμόδιου φορεί, να έρθουμε εδώ στην Επιτροπή σα και να ε, σα παρουσιάσουμε μια ανάλυση όλων των διορθωτικών και προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν σε αυτή την περίοδο. Τέλο, συμφωνούμε πλήρω ότι οι δημοσιονομικέ διορθώσει δεν μπορούν να αποτελούν αυτό σκοπό. Είναι ένα εργαλείο. Και ένα εργαλείο το οποίο αξιοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου. Άρα λοιπόν θεωρούμε πως στη νέα περίοδο 2014-2020 ε, και την παρακράτηση του 20% των πληρωμών της Επιτροπής ε, σε κάθε έτος έως τον τελικό ε, απολογισμό ο οποίος θα πρέπει να γίνεται δεκτός έως τον Μάιο κάθε χρήση, σίγουρα θα υπάρχει υψηλότερο βαθμός προστασίας του προπολογισμού στο πλαίσιο της κάθε δημοσιονομικής χρήσης. Έτσι δηλαδή οι ε, διάφορες αναστολές ε, στα προγράμματα ενδεχομένως να είναι λιγότερο αναγκαίες στο μέλλον. Αλλά όταν θα έχουμε από εκεί και μετά, ε, θα έρχομαι στη φάση τη ακαθάριση, του κλεισίματο δηλαδή το λογαριασμών, θα πρέπει να διαπιστώνουμε ποιε είναι οι δηλωτήσει δαπάνε. Εάν λοιπόν ο σχετικό κίνδυνο υπερβαίνει το 20% τη παρακράτηση από τη πλευρά τη Επιτροπή, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλαμβάνει δράση και να σταματάει την καταβολή των πληρωμών. Εάν δεν υπερβαίνει αυτό το ποσοστό, ε, το σχετικό ε, πρόβλημα και ότι το πρόγραμμα δηλαδή αξιοποιεί το 20% ε, προκειμένου να δηλώνει δαπάνες όπου υπάρχει, υπάρχει υψηλό ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να ασκεί πιέσει στα κράτη-μέλη του ώστε να σέβονται τα σχετικά συστήματα. Ε, Τέλο, αναφέρθηκε νομίζω από τον κυρία το ζήτημα του μακροπρόθεσμου αντικτύπου των λόγων προληπτικών δράσεων στα συστήματα των κρατών μελών. Νομίζω πως το ελεκτικό συνέδριο βασίστηκε εδώ σε ένα δείγμα 20 προγραμμάτων και βέβαια ήταν θεμητό να αναμένουμε ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης που έγινε πριν και μετά από το σχέδιο δράσης να αναμένουμε ότι υπήρξε ακριβώς βελτίωση των προγραμμάτων και με βάση τα όσα σας είπα πράγματι μπορεί να υπάρξει αντίκτυπο σε ένα τμήμα του προγράμματο, για παράδειγμα σε ένα διάμεσο φορέα, χωρί όμω αυτό να σημαίνει τελικά ότι υπάρχει βελτίωση σε σχέση με όλου του εμπλεκόμενου φορεί, σε σχέση με όλα τα, τις επιμέρους διαστάσεις του προγράμματο. Γι' αυτό ακριβώ θέλουμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τι ε, αρμόδιες αρχέ των κρατών μελών προκειμένου να ε, μοιραστούμε τι εμπειρίε μα και να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στο πλαίσιο ακριβώς της άσκησης της εποπτείας από πλευρά της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πρώτο και ζητώ συγγνώμη που ακρηγόρησε. Ε, Εμεί σας ευχαριστούμε για τη συνδελεχή σας απαντήσεις. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά και τώρα θα δευτερολογήσει και θα ολοκληρώσει το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστούμε Πρόεδρε όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που ανέφερε ο εισηγητής. Σας παραπέμπω στα όσα είπε η Επιτροπή ότι Προφανώ θα πρέπει οι μισοί να συρρυκνωθούν, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποια επιχειρησιακά προγράμματα. Οπότε τα συμπέρασματα που έχουμε αντιλήσει δεν ισχύουν ακριβώ όπω ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτά τα αναφέρουμε στην έκθεσή μα στην παράγραφο 106 έως την παράγραφο 110. και κατόπιν σχέση που είπε η Τλαμπατζόβα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ απορρόφησης και σφαλμάτων όσο πιο αργή η απορρόφηση πιο πολλά τα λάθη το ένα είναι συνέπεια του άλλου στην εκθεσή μας τα λέμε στην σελίδα 40 και το εξετάζουμε σε σχέση με τις δημοσιονομικές ε, ε, διορθώσεις πρόεδρος και τώρα θα δευτερολογήσει ο εισηγητής μας κύριε Πύρινσκη πολύ σύντομα πρόεδρε αυτή τη φορά ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί όσα μας είπε ήταν ε, ακριβή και ολοκληρωμένα ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου, τον κύριο Γκρέτον. Πραγματικά θεωρώ ότι όλοι μαζί θα πρέπει να επιδιώξουμε να αξιοποιούνται τα μαθήματα τα οποία λαμβάνουμε και να μην κάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη. Υπάρχει ένα σύστημα επισήμανσης, ε, κάποιο καμπανάκι όσον αφορά δηλαδή τα επαναλαμβανόμενα λάθη. Οπότε και να μην επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά οι λάθος πρακτικές. Κύριε Πυρνίκη, σας ευχαριστούμε για αυτές τις δύο εκθέσεις, τις ειδικές εκθέσεις που είχατε λέω τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ ολοκληρωμένα τα όσα μας εκθέσατε. Όμως, γιατί ε, την επόμενη έκθεση είμαι εγώ εισηγητής και όχι εσείς. Πρόκειται για το σχέδιο έκθεση για τον έλεγχο δαπανών και παρακολούθηση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων της Ένωσης. Εγγύσεις για την νεολαία. Βοήθησαν πάρα πολλοί σκιώδεις και άλλοι συνάδελφοι στην ε, Επιτροπή μας. Στο παρελθόν έχουμε συντάξει γνωμοδοτήσει όσον αφορά την ανεργία των νέων σε σχέση και με τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου την ε, τελευταία χρονιά. Και σας το λέω σε κάθε μας συνάντηση που θα συζητούμε. Νομίζω ότι η ανεργία των νέων είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του καιρού μας. Είδατε σε κάποιες χώρες τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Είναι σκανδαλώδες. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Δεν κάνουμε αρκετά για να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους. Ας κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον αυτό δεν κάνουν τα κράτη-μέλη. Ευτυχώς έχουμε βέβαια αυτό το καινούριο σύστημα των εγγύσεων για την νεολαία. Είναι σημαντική επιτυχία. πρέπει να υπάρχει front loading για την χρηματοδότηση δηλαδή να μην περιμένουμε για την εκταμείευση την ολοκλήρωση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό προσπάθησε να πετύχει το Κοινοβούλιο. Πάντως, αυτά τα μέτρα έπιασαν τόπο. Έπεσε η ενεργεία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανεργία όλων και των νέων. Νομίζω ότι βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας αυτή την προσπάθεια. Τέλος του 2016 στην Ένωση ήμασταν σχεδόν στο 19% ανεργία για τους νέους. Και αυτό φυσικά απαράδεκτο είναι, άρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Γι' αυτό και χάρηκα για αυτή την απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου να παρατείνουμε μέχρι το 2020 τουλάχιστον αυτή την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Πάντως, πρέπει να επιστρέψουμε περισσότερη πλεκοδότηση, περισσότερους πόρους. Είχαμε τα 6 δις, μετά άλλο ένα δις, όπου και τα συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο, πολλά χρήματα είναι αυτά. Αλλά φορούν όλους τους ανέργους στα 28 κρατη μελια Πρέπει να εξετάσουμε και τους ίδιους πόρους. Θα πρέπει αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσει και να το λύσει η Ένωση και τα κράτη-μέλη μαζί. Άργησαν τα κράτη-μέλη να ξεκινούν τις προσπάθειες να υλοποιούν αυτό το, το πρόγραμμα. μεταβιαστήκανε, δεν υπήρχαν σωστέ κατευθυντήριε. Τέλο πάντων γίνανε κάτι βελτιώσει και στα κρατημέλη έκαναν κάποιε μεταρρυθμίσει ώστε να εξασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση του προγράμματο. Α από άλλε εκθέσει του Ελληνικού Συνεδρίου ξέρουμε ότι δεν είχαν γίνει αρκετέ ε, συζητήσει με του εθελοντέ, με τον τριτογενή τομέα, με τι επιχειρήσει, ούτω ώστε πώ θα υπάρχουν ε, προτάσεις προσφορές θέσεων απασχόλησης προς τους νέους. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά και για την κατάρτιση ότι θα πρέπει να υπάρχουν προσφορές για ποιοτική απασχόληση στους νέους. Δεν να τους ε, προτείνουμε ό,τι να είναι. Θα πρέπει να είναι η πρόταση απασχόλησης ποιοτική. Αυτά τα έχουμε κάνει και στο παρελθόν στην Βρετανία. να Προσλαμβάνονται, ναι, και τους λένε να φτιάχνουν τον καφέ και να βγάζουν φωτοτυπίες. Ε, δεν είναι αυτή η σωστή δουλειά, ούτε τους γίνεται η σωστή κατάρτιση. Έχουν θέσεις ποιοτικέ. Έτσι θα δίνουμε ευκαιρία. Και βέβαια είναι δύσκολο να οριστεί το τι θα πει προσφορά απασχόλησης ποιοτική. Ίσως μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό η Επιτροπή. Επίσης, στο κειμενό μου αναφέρω τα των εκθέσεων για τα δεδομένα, τα διάφορα στοιχεία ή αυτό σχετίστηκε με τον προϋπολογισμό. Ε, προβληματίζεται σε σχέση με τα στοιχεία για τους δικαιούχους στο Ελληνικό Συνέδριο, τι γίνεται με τα αποτελέσματα. Ότι που είναι εμβαλωματικά τα στοιχεία που έχουμε και οι πληροφορίες. Πρέπει να είναι συμβατά τα μέτρα, τα σχεδόν πληροφορίε που μας δίνουν. Να υπάρχει μέρος συγκρισιμότητα στα στοιχεία μεταξύ των μελών. Ο καθένας άλλα μέτρα. Άρα Πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτό το μέτωπο. Επίσης, έχουμε το mismatching των, των δεξιοτήτων. Πρέπει να, να συντεριάζουν, ας πούμε. Ο καθένας δηλαδή να φροντίζει για δεξιότητες που χρειάζονται στην οικονομία του. Και έτσι είναι πιο εύκολο θα μπορούν να βρουν μια θέση απασχόλησης στο μέλλον. Πήγα να πω εδώ, τελειώνω πρόεδρε, αλλά εγώ είμαι ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή μας. Και όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, αυτό είναι σχεδικημένο. Οπότε περιμένω τα σχόλια των σχεδόν εισηγητών και των άλλων συναδελφών. Εδώ βάζω τελεία και για να δούμε τώρα. Ας λάβουν το λόγο οι σχεδόν εισηγητές. Ο κύριος Σάλα Φράγκα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. En primer lugar, quisiera eh, agradecer su trabajo sobre un tema sensible, como usted ha explicado, muy sensible para la Unión Europea. La gente joven que está. Μπράβο, μπράβο, καλά τα λέτε, γιατί eh, έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ενέργων ε, νέων. Τρομερά ποσοστά. Ενώπιν του βρισκόμαστε που από οικονομικής πλευράς είναι αφόρητο και απαράδεκτο από πολιτικής πλευράς και επίσης είναι αφόρητο και από πλευράς ηθικής. Άρα χρειάζεται τώρα να αναλύσουμε το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα πετύχει με την εγγύηση για την νεολαία και νομίζω ότι βέβαια οι υπερκοδοτήσεις είναι πολύ σημαντικές οικονομικά και καλά τα λέει ναι, στην εκθεσή σα ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον χώρο αυτών των νέων. Στου νέου δηλαδή πού είναι, πού, πού δουλεύουν και πού σπουδάζουν και κατά πόσον πραγματικά αναφέρονται, συγγνώμη, ε, ενδιαφέρονται να αναζητήσουν θέση εργασία. Όλα αυτά είναι σημαντικό πρόεδρε. Επίσης το να μπορέσουμε να πετύχουμε αρμονία να δουλεύουμε συντονισμένα με τα κρατημέλη. Δεν ξέρω αν το θέμα αυτό είναι αποκλειστικά δημιουργικό. Γιατί υπάρχουν κρατημέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα 100% κάνει όσο πρέπει να κάνουν πλευρά προπολογισμού. Γιατί αυτός ο κανονισμός, αυτό το πρόγραμμα προσφέρει περισσότερα που δεν τα έχουν εκμεταλλευτεί. Άρα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, να υποπτεύσουμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει και εμείς και η Επιτροπή να προσέξουμε και να τοποθετηθούμε με κρυστάλλινες θέσεις. Όπως είπατε και έχουμε διαφοροποιημένες αντιδράσεις. Όμως, σχεδόν κατά 7 μονάδες έπεσε η ανεργία. Αλλά έτσι κι αλλιώς οι επιδόσεις μας δεν μας κολακεύουν. Να προσπαθήσουμε να ρίξουμε και άλλο την ανεργία. Εμείς από πλευρά ΕΛΚ είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε για την εκθεσή σας. Νομίζω ότι όσα αναφέρονται είναι λογικά και γενικά συμφωνούμε με το κείμενο. Έχουμε Κάποιε προτάσεις τροπολογιών, δεν επηρεάζουν την ουσία του κειμένου σας, απλώς θα πρέπει να δούμε για το πώ θα συμφωνήσουμε στο πώ θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε τι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε ω πόρου τι θα πρέπει να μετέλθουμε ούτως ώστε αυτοί οι που θα διατεθούν να είναι αποτελεσματικοί πρόκειται για κορυφαία προτεραιότητα της Ένωσης ε, σε αυτό το σημείο συμφωνούμε με όσα λέτε κύριε Σιγητά και σας ευχαριστώ ως πρόεδρο εγώ ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας περιμένω τις τροπολογίες σας λέει ο πρόεδρος Μαρτίνα έχεις το λόγο Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε μπορώ να μιλώ για ώρες για το θέμα αυτό με ενδιαφέρει πολύ θα περιστώ σε ορισμένα μόνο σχόλια διότι βεβαίω ε, έχουμε ήδη συζητήσει για το θέμα αυτό, αλλά η συζήτηση ήταν διαφορετική. Ευχαριστώ για την δουλειά που κάνατε. Νομίζω ότι έχετε όντω θίξει τα πιο σημαντικά θέματα. Θέλω να δώσω κάποια έμφαση σε ορισμένα πράγματα. Όπω είπα και στην Επιτροπή Απασχολήσεω και πρώτα βέβαια η οικονομική αποδοτικότητα που δεν είναι ειδικά για την απασχόληση αλλά μακροπρόθεσμη απασχόληση, απόκτηση προσόντων που να ζητούνται από την αγορά εργασίας και πρέπει να είμαστε προσεκτικές να μην θεωρήσουμε αποτελεσματική κάποια προσφορά η οποία είναι ad hoc, είναι επί τούτο. Η εφαρμογή της εγγύησης ε, νεότητας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη, διότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε την προσπάθεια επιλύσεως των προβλημάτων, αλλά και αποτελεσματικά ταυτόχρονα. Επομένω να λάβουμε υπόψη τη ανάγκες τη αγορά, αλλά να χορηγήσουμε κατάρτιση, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση. Η πιο μεγάλη συζήτηση στην Επιτροπή Απασχολήσεως ήταν αυτό που είπατε κι εσείς, δηλαδή προσφορά ποιότητας. Πώς ορίζεται η προσφορά ποιότητας, γιατί όσο γνωρίζετε και ω φιλελεύθερο, πρέπει να είναι διαφορετική η ποιότητα της ε, προσφοράς κατάρτισης ανάλογα με την χώρα, αλλιώ στην Ισπανία, αλλιώ στην Τσεχική Δημοκρατία, αλλιώ για τον ένα, αλλιώ για τον άλλο. Πάντω χρειάζεται κάποια αφετηρία, κάποια αρχή ενό ορισμού. Και ο ορισμό, μια καλή βάση για τον ορισμό που βρήκαμε στην Επιτροπή Απασχολήσεω είναι προσφορέ θεωρούνται καλή ποιότητα εφόσον βοηθούν να συντεριάξει το προφίλ του ενδιαφερομένου, ανάγκε τη αγορά και η μακροπρόθεσμη απασχόλησή του στην αγορά εργασία. Είναι καλή αφετηρία αυτή, αλλά βέβαια κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη δική μα πρόταση δηλαδή τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολισμού δεν αρκεί, διότι δεν είναι μετρήσιμο ο ορισμό αυτό. Δεν μπορεί να μετρήσει κανεί με πραγματικού δείκτε. Ε, ήταν κάπω ακαθόδε αυτό. Επίσης, η ανάπτυξη, δηλαδή τέλο πάντων η προσπάθεια ε, δημιουργής ορισμού δεν εγγυάται την θετική εφαρμογή της, ε, της ε, εγγύησης για νότητα. Από την άποψη της Επιτροπής Απασχολήσεως έχουν γίνει ορισμένες προτάσεις για την ηλικία των συμμετοχόντων ότι θα πρέπει δηλαδή, το όριο να φτάσει στα 30 έτη ηλικία. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή θεωρώ 25 χρόνια της ηλικίας είναι σωστά, γιατί είναι και η πιο ευάλωτη ας πούμε, ηλικία των νέων. Είναι κάτι όμως που πρέπει να συζητηθεί στο μέλλον, όντως. Για να ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι η χρηματοδότηση δεν αρκεί. Χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες μέλη. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις απαιτούνται πράγματι και στις αγορές εργασίας αλλά και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Πρέπει να ενισχυθούν οι διοικητικές ικανότητες των χωρών μελών. Το είδαμε αυτό και πέρσι όταν πήγαμε στην Καλαβρία και στην Σικελία της Ιταλίας για να δούμε την εφαρμογή της εγγύης νότητας και διαπιστώσαμε πλήστα προβλήματα ε, διοικητικής ικανότητας. Χρειάζεται και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Ευρωπαϊκό επίπεδο, εθνικό, περιφερειακό. Αυτό αυτές αδυναμίε διαπιστώσαμε στην Ιταλία. Και είναι κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να περιληφθεί στην έκθεσή μα. Η σημασία δηλαδή τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβερνήσεω. Και τελευταίο, και σα ευχαριστώ που το θέσατε, η έλλειψη συντέριαξη, ας το πω έτσι, των ε, προσόντων. Την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Απασχολήσεω ενέκρινε την έκθεσή μου για το ίδιο θέμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τα προσόντα, τις δεξιότητες για το μέλλον. Και κάτι που χρειάζεται ακόμη είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται να λησμονούμε. Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε στην παρούσα επιτροπή. Το μόνο σημείο στο οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε είναι η cost effectiveness, η αποδοτική χρήση δηλαδή των πόρων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλλη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα για την ανεργία των νέων, ιδίως όσον αφορά στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, γιατί εκεί ο κόσμος είναι πιο στριμωγμένος, εκεί πάνω πιο σημαντικές ε, ανισορροπίες. Ε, θα πρέπει να ξεβρεθούν κάποιε λύσεις και ελπίζουμε σύντομα, άντε να γίνουν εκλογές στην ε, Γερμανία, ούτως ώστε να δούμε καμία αλλαγή. Δεν το πολύ πιστεύω εγώ. Είπαμε είναι σημαντικά τα νούμερα όσον αφορά την ενεργεία των νέων. Και βέβαια χρειάζεται να κάνει περισσότερη προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ με αυτά που προτείνατε γιατί και στη χώρα μου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει διοικητικά, να δοθούν οδηγίε κατευθυντήρε, τι να κάνουν οι αρχές για να διαχειριστούν το πρόβλημα ε, από πλευρέ διοικητικέ, αλλά θα πρέπει να πληρώνονται βέβαια ναι, ε, γιατί όπω είπε το ελληνικό συνέδριο ε, πολλές φορές βρίσκουν δουλειά κάποια θέση εργασία, αλλά βάζουν λεφτά από την τσέπη του. ζουν από τα δικά τους λεφτά γιατί για ένα μεγάλο διάστημα δεν του πληρώνουν αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Και επομένως θα πρέπει να λάβουμε σκληρά, αυστηρά μέτρα και να μπορέσουμε να τους δώσουμε ποιοτική απασχόληση. Και έτσι, να, με κάποιους τρόπους τέλος πάντων να αυξηθεί η ζήτηση για εργαζομένους, για εργαζομένους σε θέσεις ποιοτικέ και να δούμε το ότι εάν δεν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση, εάν δεν υπάρχει κάποιο είδου σχεδιασμό, εάν δεν επικεντρώσουμε την προσοχή μα βουλά πολιτική, εκεί που πρέπει, είναι πολύ δύσκολο να τονώσουμε την ζήτηση για θέση απασχόληση. Δύσκολα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει σε αυτό τον ε, στόχο. όπως το έχουμε ξαναβεί ως πολιτική ομάδα. Επιμένουμε ότι χρειάζεται να αναθεωρηθεί το πλαίσιο διακυβέρνηση που έχουμε και έτσι να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχουν, να τονώσουν την ζήτηση. Γιατί εάν το κάνουμε αυτό, όλα αυτά τα διοικητικά προγράμματα, αυτές οι εγγυήσεις για την ανεργία των νέων όλα αυτά τα σχετικά προβλήματα όλων αυτών που ψάχνουν δουλειά δεν θα γίνει τίποτα εάν δεν έχουμε αύξηση της συζήτηση, αναθέρμανση της οικονομίας χτυπήσουμε την ανεργία και έτσι αυτά είναι οι βασικές μας παρατηρήσεις Thank you. Uh, next speaker, Ευχαριστούμε. Κύριο Σέπιρινς και ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και συμμερίζομαι βασικό σκεπτικό, αν θέλετε, συλλογιστική της έκθεσής σας και συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο ως προς την ε, διαπίστωση που έκανε ως προς την απαράδεκτη κατάσταση που έχουμε σε μία σειρά από ό,τι αφορά την ανεργία των νέων. Ε, θα ήθελα όμως να τονίσω μία ιδιαίτερη πτυχή που αξίζει εδώ να αναφερθεί το ότι δηλαδή κάποια κράτη-μέλη ξεκίνησαν κάπως, κάπως αργοπορημένα στις προσπάθειες τους. Δηλαδή ακούμε ε, συνέχεια ότι υπάρχουν χρήματα που ταπανώνται χωρίς όμως να βλέπουμε τα αποτελέσματα και η έκθεση ε, που είχαμε δει και η οποία χρησιμοποιούσε ε, δεδομένα από το 2015 ήταν αρκετά απογοητευτική. Κάτι λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι τα συστήματα αυτά έχουν δημιουργηθεί αφενός για να δημιουργούν θέσεις εργασίας, αλλά αφετέρου για να δημιουργούν συστήματα, δομές στα κράτη-μέλη, μέσω των οποίων θα είναι ε, πολύ ευκολότερο να, να αναγνωρίζονται τα κοινωνικά, αν θέλετε, στρώματα όπου οι νέοι ακτίβως βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και προκειμένου να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα όπου οι εν λόγω νέοι δεν ε, αναβρίσκουν θέσεις μαθητείας ή απασχόλησης που δεν είναι αρκούντως ε, ενδιαφέρουσες. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε και όταν εξετάζουμε το ζήτημα της σχέσης κόστους αποτελέσματος αυτών των συστημάτων της εγγύησης για την ενολέα, θα πρέπει να αξιολογούμε και αυτή την πτυχή, κατά πόσο δηλαδή δημιουργούν αυτές τις ικανότητες, δημιουργούν αυτές τις δομές στα κράτη-μέλη και πόσο, σε ποιο βαθμό έχουν βελτιώσει τη ε, τη, τη, τη, λειτουργία αυτών των συστημάτων ακριβώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τι ενόχο προκλήσει. Δηλαδή, δημιουργία θέσεων εργασία, ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν ή να, να ε, αποτέχονται θέσει εργασία και ούτω καθεξή. Και κάτι ακόμα που ανέφερε και ο κ. Ε, Μαρκιάλη είναι ότι υπάρχει και μια οριζόντια διάσταση του προβλήματος. Δηλαδή, οι σχετικέ εγγυήσει ε, και η εγγύηση ιδιαίτερα για τον έχει ένα γενικότερο χαρακτήρα, δηλαδή έχει ε, όμως από εκεί και μετά να κάνει για παράδειγμα με, τους, ε, με τον, ε, ένα πιο περιφερειακό χαρακτήρα, δηλαδή για παράδειγμα ε, περιοχές στις οποίες είναι λιγότερο λογιστικές οι θέσεις εργασίας και εδώ έχουμε να κάνουμε και πάλι με τις ε, περιφερειακές, με την περιφερειακή ανάπτυξη και τα σχετικά προγράμματα. Εδώ έχουμε πάλι να κάνουμε και με ε, περαιτέρω πρωτοβουλίες γιατί Ε, ουσιαστικά ε, κατηγορείται η πρωτοβουλία ε, αυτή για την ανεργία των νέων ως συμπέστηνη αν θέλετε για την γενικότερη ανεργία. Σίγουρα θα πρέπει να αξιολογούμε τέτοιου είδους προγράμματα από την δημοσιονομική άποψη, αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να τα θεωρούμε ως την πανάκια για την επιλύση των σχετικών προβλημάτων. Πιο πολύ θα πρέπει να θεωρούνται δηλαδή ως η αιχμή του δόρατο τη όλη προσπάθεια ε, που γίνεται για αντιμετώπιση του, πρόβλημα, του προβλήματος. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Ο Μπράιν έχει το λόγο. Ναι, θέλουμε και εμεί να ευχαριστήσουμε για αυτή την έκθεση και νομίζω πω ε, υπάρχει μια γενικότερη υποστήριξη από τι πολιτικέ ομάδε απέναντι στην ε, δουλειά που κάνετε. Δηλαδή, ε, ακόμα κι αν αλλάζουμε λίγο την έμφαση που δίνουμε και πάντοτε έχουμε έναν ίδιο στόχο. Και όπω είπε πολύ σωστά ο κύριο Πυρίνσκης, θα πρέπει από τη μία πλευρά να εξετάζουμε κατά πόσο έχει πράγματι αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η χρηματοδότηση εδώ προκειμένου να αντιμετωπιστεί σκανδαλώδης πραγματικά σε ορισμένα κράτη-μέλη κατάσταση ό,τι αφορά την ανεργία των νέων. Αλλά από εκεί και μετά ο στόχο είναι και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ακριβώ να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη για να δημιουργήσουν καλύτερα βελτιωμένα συστήματα. Και είναι ενδιαφέρον ε, να διαπιστώνουμε όπου ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία ε, ιστορικά έχουν καλύτερες θέσεις με σε κατάρτιση κατάρτισης ε, και όπου υπάρχει και χρηματοδότηση αυτών των θέσεων από τα κράτη-μέλη υπάρχει και πολύ χαμηλότερα, χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, εγγύηση για τους νέους εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με την μείωση τη ανεργία των νέων που πραγματικά είναι απαράδεκτα υψηλή αλλά έχει να κάνει και ε, με το πώ αξιοποιούμε καλύτερα αυτέ τι ε, θέσει μαθητέ, πώ ε, αξιοποιούμε αποτελεσματικότερα τα κοντιλιά μα, πώ μαθαίνουμε καλύτερα ο ένας από τον άλλον για παράδειγμα να δώσουμε μια απάντηση ω προ το κατά πόσο είναι καλύτερο να λαμβάνει κανεί πανεπιστημιακού τύπου εκπαίδευση αν είναι καλύτερο να έχει μια πρακτική εξάσκηση σε μια πραγματική θέση επαγγελματή κατά τη μαθητείας και από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποιε αγορέ εργασία, οι οποίε πιο ε, αποτελεσματικέ στη λειτουργία του, οι οποίε είναι πιο διεθνοποιημένε. Και έτσι θα πρέπει να δώσουμε τις ε, σχετικά, τα σχετικά ενάπτυσματα ε, στου ε, συμμετέχοντε για να, για να μπουν σε αυτήν την ε, αγορά εργασία. Για παράδειγμα, εγώ προέρχομαι από το Δουβλίνο, έχουμε μια πολύ διεθνοποιημένη αγορά εργασία. Δηλαδή, έχουμε διάφορου συμμετέχοντε σε αυτή την αγορά, ενδιαφερόμενου για αυτή την αγορά και έτσι τα, στα κράτη-μέλη εκείνα, στα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί εν λόγω ευκαιρίε, θα πρέπει να προωθήσουμε το, το σχετικό οικονομικό μοντέλο τη αγορά εργασία. Από εκεί και μετά, όπω σωστά αναφέρετε στην έκθεσή σα και αναφέρετε προκαταρκτικά, έχει σημειωθεί πρόοδο. Όμω, ε, πραγματικά παραμένει απαραδεκτό υψηλό το, υψηλό το ποσοστό της ανεργίας των νέων στο 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω πως ε, τα όσα έχουν συμβεί στο επίπεδο των οικονομιών μας ε, κατά τα τελευταία τρία χρόνια στην Ευρωζώνη ε, είναι θετικά. Δηλαδή, παρότι έχουμε θετικέ εξελίξει στη γενικότερη οικονομία τη Ευρωζώνη, πολλοί νέοι μα δεν έχουν δει κάποιον αντικτύπο στη ζωή του. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση για να επωφεληθούν και εκείνοι. Οπότε, σωστά λέτε, Πρόεδρε, χρειαζόμαστε δεδομένα εδώ, περισσότερα δεδομένα. Καλά παραδείγματα, κακά παραδείγματα και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη τα οποία είτε κινούνται αργά, είτε δεν έχουν δημιουργήσει ένα βιώσιμο μοντέλο τη αγορά-εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη αυτά να βελτιώσουν τι επιδόσει του. Και τέλο, να πω ότι υπάρχει σχέση μεταξύ υψηλών ε, θέσεων εργασία ε, στην αγορά, υψηλού αριθμού θέσεων εργασία στην αγορά και φορολόγηση, επίπεδου φορολόγηση. Αυτό δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, εάν φορολογούμε ε, πάρα πολύ εξοντωτικά, αν θέλετε, του νέου μα σε ένα κράτο μέλο, τότε εν λόγω ε, νέοι θα ε, αναζητήσουν εργασία σε άλλο κράτο μέλο. Οπότε υπάρχει σχέση μεταξύ υψηλού ποσοστού ανεργία αφενό και υψηλή φορολογήση αφετέρου. Και ε, για παράδειγμα, ένα ποσοστό τη τάξη του 12 15% σε φορέ είναι ένα παράδειγμα που έχουν ακολουθήσει κάποιε ε, από τι πιο προηγούμενε χώρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ακούσαμε από του ε, διάφορου συναδέλφου. Μπορούμε να ακούσουμε και από την Επιτροπή όμω ο κύριο Πιέτα Αντώνιο από τη Γενική Διεθνή Απασχόληση. Έχετε το λόγο. Ναι, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σωστά προφέρατε το όνομά μου. Καλησπέρα σε όλους και καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω ε, θερμά τον ε, συγητή, τον Βόχαν, για αυτό το σχέδιο έκθεση. Να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις συγητές και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν στη συζήτηση. Για την... Ε, γιατί βέβαια έχουμε να κάνουμε μια συζήτηση που ενδιαφέρει πολύ την, την γνώμη, αλλά και ένα ζήτημα που αφορά πολύ την Επιτροπή, δηλαδή αυτή η πρόκληση της ανεργίας των νέων. και το γεγονός ότι δηλαδή με την ε, πρωτοβουλία ε, ε, για την ανεργία των νέων δεν επιλύουμε το ζήτημα της ανεργίας των νέων και ότι χρειαζόμαστε μια πιο ολιστική προσέγγιση όπως πολλοί από σας αναφέρατε. Υπάρχουν κάποια, κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις, για παράδειγμα από το 2014 16 εκατομμύρια νέοι έχουν συμμετάσχει σε συστήματα εγγύηση για τον νέο και 10 εκατομμύρια έχουν λάβει θέσεις απασχόλησης, επαγγελματική κατάρτισης, μαθητείας ή διαβίου κατάρτιση. Από εκεί και μετά, εμ, όπως ανέφερε και το ελεγκτικό συνέδριο, ε, έχουν ξεκινήσει με κάποια καθυστέρηση εν λόγω προσπάθειε. Αναφέρετε και εσεί ε, στην έκθεσή σας τις ε, καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία, ε, η οποία οφείλεται εν μέρη στην, ε, στον διορισμό των αρμοδιών αρχών από τα κράτη-μέλη, αλλά και εδώ ουσιαστικά έχουμε ολοκληρώσει την λόγω διαδικασία, γιατί δύο κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα δηλώσει τις αρμόδιες αρχές τους. Δηλαδή 32 από τις συνολικά 34 αρμόδιες αρχές ήδη έχουν καθοριστεί. Τώρα αν δούμε τα δεδομένα από τον Ιούλιο του 2016, ένα 4,1 εκατομμύρια νέοι έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία. Ενώ το Νοέμβριο του ίδιου έτους βρισκόμαστε στο 1,6 εκατομμύρια. Οπότε δηλαδή είδαμε εδώ μια ε, μεγάλη αύξηση σε λίγους μήνες. Ε, και τώρα με την αιτήσια έκθεση εκτέλεσης ε, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό ε, Κοινωνικό Ταμείο και, την, και τις πρωτοβουλίες απασχόλησης θα δούμε και περισσότερα δεδομένα και εκεί αναμένουμε ακόμα υψηλότερε αυξήσεις σε ό,τι αφορά δηλαδή, τον αριθμό των καλυπτωμένων νέων. Τώρα, συμφωνούμε και εμείς με την έκθεσή σας, Πρόεδρε, αλλά και με την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, το ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες επαφές με τους νέους σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους. Δηλαδή έχουμε από τη μία ε, πλευρά ε, την αργία των νέων αυτή καθεαυτή και από εκεί και μετά τις ανάγκες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, πρέπει να έχουμε καλύτερους δείκτες ε, και πρέπει να παρακολουθούμε καλύτερα την όλη κατάσταση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν εδώ να υποστηρίζουμε στο βαθμό που μπορούμε τα κράτη-μέλη, είτε χρηματοδοτικά, είτε με συμβουλευτικέ υπηρεσίε ό,τι αφορά την πολιτική του, είτε με τεχνική αρρωγή επί τόπου όπου αυτό είναι απαραίτητο. Και Έχουμε επίσης ε, ζητήσει από τα κράτη-μέλη να έχουν πιο στοχευμένες προσεγγίσεις τους και να μας αναφέρουν πιο συγκεκριμένα τις ομάδες στόχους ε, των συστημάτων ε, της πρωτοβουλίας ε, της, ε, για τους νέους. Και πάντως σε αυτό το επίπεδο έχουμε θετικές ενδείξεις, δηλαδή το 2015 σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών Ε, το ίμιση όσων συμμετείχαν στο, σε αυτό το σύστημα της εγγύησης για τους νέους ήταν νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης, NEETs όπως λέγονται. Ε, επιχαίρουμε το γεγονός από την πλευρά της Επιτροπής ότι οι συνομοθέτες αποφάσισαν όχι μόνο να αυξήσουν την πρωτοβουλία, ε, να αυξήσουν τον προπολογισμό της πρωτοβουλίας κατά ένα δισεκατομμύριο, αλλά κινήθηκαν και πέραν αυτού. Γιατί συμφώνησαν τελικά σε αύξηση ύψου 2, 1,2. Τώρα, επαρκεί αυτή η αύξηση. Αυτό ήταν και το ερώτημα που έθεσε το ελεκτικό συνέδριο. Ναι, γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν επαρκεί. Γνωρίζουμε πως ε, και η Eurofound και ο ILO εκτιμούν πως η ανάγκη της επένδυσης ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση είναι πολύ ψηλότερη. Αλλά όπως ε, είπατε και εσείς προηγουμένως, η ε, λόγω πρόκληση είναι πολυδιάστατη. Οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα για να την αντιμετωπίσουμε. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ και τα εργαλεία τη οικονομική διακυβέρνηση αλλά και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και εδώ περνάω στο άλλο ζήτημα που θίξατε, δηλαδή της ποιότητας. Ποιότητας των θέσεων εργασίας, των θέσεων απασχόλησης που προβλέπονται στο πλαίσιο της εγγύησης. Εδώ λοιπόν συνεργαζόμαστε τον ε, Παγκοσμίου Οργανισμό Εργασία. και εξετάζουμε τη βιβλιογραφία, αν θέλετε, που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασία. Για παράδειγμα, με βάση τον ΩΣΑ υπάρχουν τρεις κατηγορίες, ε, ε, δηλαδή η ποιότητα των εσόδων, ύψος της ασφάλειας, αν θέλετε, δηλαδή ασφάλεια στη θέση εργασίας και εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή ωράριο εργασία και ούτω καθεξής. Η κυρία Σαββαλό πρότεινε επίση τη συμπερίληψη τη διάσταση τη βιωσιμότητα. Ε, πέραν δηλαδή τη εγγύηση σε γενικότερο επίπεδο. Όλα λοιπόν αυτά αποτελούν βήμα για σκέψη και θα τα λάβουμε υπόψη μα και μετά από την ε, πρόσκληση που μα έκανε η ΕΠΣΚΟ θα συνεργαστούμε με αυτού του διεθνεί οργανισμού αλλά και με την ΕΜΚΟ την Επιτροπή λοιπόν ΕΜΚΟ του Συμβουλίου προκειμένου να αξιολογήσουμε και να μπορούμε να αξιολογούμε τι ακριβώς, ε, ε, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα την ε, εγγύηση για τους νέους και πώς μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα την εκτέλεση των σχετικών πρωτοβουλειών. Την εγγύηση δηλαδή και την πρωτοβουλία για την αργία των νέων. Αυτά από και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θεωρώ ότι ήταν το, οποίο, το γεγονός ότι αναφέρεται ότι έχει, υπάρχει, έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά υπάρχουν και κάποια εκρεμή ζητήματα και ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εκκρεμή ζητήματα. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο τώρα της έκθεσής μας νομίζω πως ε, υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ των ε, συναδέλφων ότι δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες διοικητικές ικανότητες, δομές στα κράτη-μέλη προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά το, ε, η εγγύηση για τους νέους. Νομίζω πως υπάρχουν κάποια ακόμα ζητήματα ε, επί των οποίων θα πρέπει να συζητήσουμε, όπως για παράδειγμα ε, να αποφεύγουμε την ανταδυστυχία σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικέ δεξιότητες, το ζήτημα που ανέφερε η Ματίνα, το ζήτημα της ποιότητας, ποιότητας δηλαδή της προσφερόμενης θέσης. Πρόκειται λοιπόν για εκκρεμότητε, εδώ που ακόμα θα πρέπει να ε, διορθώσουμε για ζητήματα που πρέπει να διορθώσουμε και αναμένουμε ενδιαφέρον τι ε, τροπολογίε των συναδέλφων. Για να πω εδώ ότι η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών είναι 10 Ιουλίου. Κλείνω με αυτό το ζήτημα. Αυτό ήταν το θέμα υπαριθμών 5 και πάμε στο 6 που είναι η αποστολή της Επιτροπής μας σε Κροατία και Σερβία 17 με 20 Ιουλίου το σέντρος. Έχουμε το σχέδιο προγράμματος για την αποστολή. Έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν. Είχαμε στο παρελθόν, συμπληρωθήκαν και άλλοι για αυτή την αποστολή μας σε Σερβία και Κροατία. Οπότε θα πρέπει να κλείσουμε τα εισιτήρια του αεροπλάνου όσο γίνεται πιο Άρα και πρέπει να δούμε τι λεπτομέρειε του προγράμματο. Ο σκοπό αυτή τη αποστολή είναι να δούμε τι γίνεται με την απορρόφηση των κοινωτικών πόρων σε αυτά τα δύο κράτη-μέλη. Και θα πρέπει επίση να βοηθήσουμε όσον αφορά τα διοικητικά. Βέβαια η Κροατία είναι κράτο μέλο και η Σερβία βρίσκεται στην πρωταξιακή φάση. Άρα είναι σημαντικό θα ήταν αποστολή να δούμε τι γίνεται με κάποια έργα και να συζητήσουμε για κάποια άλλα θέματα, συναντήσεις δηλαδή, με την ε, διοίκηση, με την ε, κυβέρνηση. Αν δείτε και το πρόγραμμα, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε συναντήσεις που αφορούν όλα αυτά που σας είπα. Όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει το πρόγραμμα τώρα. Ε, έχουμε όμως και προσώπους Επιτροπής, οι οποίοι και αυτοί ίσως θέλουν να λάβουν το λόγο. για τη Σερβία. Έχουμε ένα τάρχη. Ποιος είναι η κυρία Κάθριν Γουέντ. Και την Κροατία είναι η κυρία Νιρβάνα Μπίσιβιτς. Είστε εδώ. Α, μάλιστα. Οπότε ίσως μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά αυτές τις χώρες. Αυτά θα μας είναι χρήσιμα σε αυτή την ε, επιστολή, αποστολή του Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να σας τα πω εγώ πρώτη, γιατί θα αρχίσετε από τη Σερβία. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τη διαδικασία της προσχώρησης της Σερβίας, να δούμε και την πολιτική συγκυρία. Πριν πάμε στα θέματα της αρρωγής προς τη χώρα, η πολιτική συγκυρία χαρακτηρίζεται από κάποιες ε, πρόσφατες αλλαγές, αλλά και από σταθερότητα είχαμε εκλογές το 16 και φέτος τον Απρίλιο είχαμε προεδρικές εκλογές όπως προβλεπόταν κατέβηκε ο πρόεδρος και ξανακέρδισε το αξίωμα του πρόεδρου όλα ήταν καλά οργανωμένα αλλά ο ΣΑ ε, επικρίνει την εκλογή διαδικασία και λέει ότι υπήρχε ένα κλίμα από τον τύπο, από την κυβέρνηση και ότι κάτι χράστη τη του το κυβερνούν κόμμα όσον αφορά τι εκλογέ. Όπω είπαμε, ο πρώην Πρωθυπουργό 1η Ιουνίου ανανέωσε την εντολή του ε, και έγινε πρόεδρο, οπότε θα σχηματίσει κυβέρνηση τέλο του μηνό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, θα έχουμε ένα νέο Πρωθυπουργό επομένω, που θα οριστεί, θα επικυρώσει το Κοινοβούλιο την εκλογή του και θα είναι γυναίκα για πρώτη φορά στη χώρα. Ο νέος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι οικικό στόχο της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι αυτό είναι προτεραιότητα και για να δούμε τώρα τις διαπραγματεύσεις προενταξιακέ. προενταξιακές είπαμε ότι έχει σταθερή ρότα η χώρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όπως ας πούμε στο ε, Μαύρο Βούνιο 73% είναι ο κόσμος ε, υπέρ ε, και πολύ λιγότερο στη Σερβία. Ε, υπάρχει σημαντική επιρροή και παρουσία στα μέσα της χώρας και στην πολιτική ζωή σκιά της Ρωσίας. Ε, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ένταξη της χώρας. Βέβαια η χώρα είναι πολύ δραστήρια, και διαπραγματεύσει έχει 10 κεφάλαια. Είχαμε διακυβερνητική συνάντηση πριν εβδομάδα και ίσως σας ενδιαφέρει σας. Οι Σέρβοι λένε ότι η διαδικασία προχωράει αργά. Θα ήθελα να ανοίγουν και να κλείνουν τα κεφάλαια πολύ ταχύτερα. Από πλευρά Κομισιόν κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς για να κινηθούμε ταχαίως. Ε, για αυτή τη διαδικασία έχουμε επαφές με τη διοίκηση της χώρας, με τους διαπραγματευτέ που τους βοηθούμε να προχωρήσουν και αυτοί και θα μπορούσαμε να ανοίξουμε και άλλα κεφάλαια κατά την επόμενη Εστονική Προεδρία. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τη Σερβία. Καταρχήν είναι θέμα τη θεματολογία του μεταρρυθμιστικού της χώρας ε, ρίος το κράτος δικαίου, μεταρρύθμιση της διοίκησης και οικονομική διακυβέρνηση. Έχουμε τώρα δύο τομείς όπου ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων διακυμαίνεται γιατί το θέμα είναι το κράτος δικαίου και ο διάλογος με την Πρίστινα. Οπότε εμείς Έχουμε την υπηρεσία μας εκεί και υποβάλλει έκθεση κάθε εξάμεινο για το αν εξαμαλύνονται τα πράγματα, τι γίνεται το κράτος δικαίου. Πάντως υπάρχει πρόοδος και ας μην είναι τόσο ταχεία. Δεν μπλοκάρονται επομένω τα σχετικά κεφάλαια της διαπραγμάτευσης. Για να δούμε τώρα για την ε, βοήθεια προς τη χώρα, την χρηματοοικονομική ενίσχυση, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δίνουμε στη χώρα μέσω του σχετικού οργάνου ε, του προενταξιακού για μεταρρυθμίσεις για την όλη διαδικασία ένταξης διακυβέρνηση, δικαιώματα, ενέργεια, κράτος δικαίου, μεταφορές, περιβάλλον, ανταγωνιστικότητα, γεωργία κλπ. Και σύμφωνα με αυτά που ισχύουν κάθε χρόνο καλύπτουν στον προγραμματισμό κάποιου τομεί τη οικονομία, ούτω ώστε να μπορούμε να πιάσουμε όσα κάνουμε περισσότερο τόπο και όλα αυτά είναι σημαντικά για την ένταξη της χώρας και κάθε φορά που θα με αυτή η τομή κάθε φορά πόσο όροι μείνει τι γίνεται. Τώρα τώρα κοιτούμε τα χρηματοοικονομικά και θα δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση. Αυτά τα προγράμματα, τα έργα που θα δείτε αφορούν κάποια προγράμματα του 12 και του 13. Τότε ο χρόνος πιέζει λιγότερο, τώρα πιέζει περισσότερο για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, τώρα για τα έργα υποδομής. Ε, βοηθούμε την ε, χώρα και, και έχει ε, κάποια τέτοια έργα και προγράμματα για τα έργα υποδομής τα που χρηματοδοτούμε εμείς ή χρηματοδοτούνται από διάφορα εθνικά ταμεία και όσον αφορά την έμεση διαχείριση, το 13 για πρώτη φορά ανέλαβε τη διαχείριση η χώρα των κοινωτικών πόρων, γιατί θεωρήσαμε ότι μπορεί η χώρα να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα. Οπότε, το 2014 επίσης είχαμε αυτοδιαχείριση ας πούμε και αποφάσισε το 2014 η Επιτροπή να εστιάσει ε, αυτή την ε, ρύθμιση της έμεσης διαχείρισης και σε διάφορα έργα, προγράμματα για περιβάλλον, ενέργεια, αυτά τα είπα, τους, αυτούς, αυτή την πολιτική αφού και τη γεωργία και η πρώτη πρόκληση για τη χώρα για την άμεση διαχείριση ήταν το 2013 και είχαμε τότε μια προθεσμία που τέθηκε για αυτό τον μήνα και πήγαμε σε 85% απορροφητικότητα και απορρόφηση πολύ σημαντικό λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν κατά τη σύναψη της συμφωνίας όσον αφορά το προσωπικό και όσον αφορά τα του οικονομικού ελέγχου. Άρα όλα αυτά είχαν δημιουργική αντιμετώπιση. Θα πάτε και θα δείτε τι γίνεται όσον αφορά τη δημιουργία δυνατοτήτων και όσον αφορά την τεχνική αρρωγή προς τις αρχές της χώρας για την διαχείριση της βοηθείας. Όλα αυτά κάνουμε για να πλησιώσουμε του θεσμούς τη χώρα. Αντλήθηκαν κάποια συμπεράσματα από τον πρώτο κύκλο προσπαθειών για να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον, στα πρόγραμματα που θα ακολουθήσουν. Επίστευουμε ότι είναι σημαντικό το πώ θα βελτιώσουμε το, με σύστημα, να υπάρχει υγιής διαχείριση των οικονομικών για ό, όλους τους πόρους αυτούς και γι' αυτό και έχουμε το κεφάλαιο 32 του χρηματοοικονομικού ελέγχου. Η Σερβία έχει ένα σύστημα μεταρρύθμισης το εγκρίνει τον Δεκέμβριο του 2015 ε, έχουν λάβει σχετικές υποχρεώσεις στο κεφάλαιο 32 των διαπραγματεύσεων και θα επισκεφθείτε ένα έργο και αφορά ε, αυτό το πρόγραμμα τη βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών και αυτό το έργο που θα δείτε ε, αφορά 80 εκατομμύρια ευρώ ενίσχυσης. Επίσης έχουμε χρηματοδότηση για αυτή την πολιτική μεταρρύθμιση, για ανταγωνιστικότητα, για υποστήριξη των ε, ΜΜΕ, βοήθεια προς τις αρχές, ε, για την άμεση διαχείριση των κοινωνικών πόρων και εν κατακλείδη να σας πω κάτι εδώ αφορά την προβολή η προβολή μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή εκεί είναι πολύ σημαντική προβολή και της Ένωσης και των κοινωτικών πόρων. Είμαστε ο πρώτος εταίρος της χώρας. Αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στα όσα δηλώνουν, στα όσα πιστεύει εκεί ο κόσμος. Θεωρούν ότι η πιο μεγάλη, τους, πιο σπουδαία εταίρη είναι η Κίνα και η Ρωσία. Άρα τα γκάλωπ δεν κατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Οπότε γι' αυτό και συνέχεια προσπαθούμε να προβάλλουμε περισσότερο το έργο μας. Και τον ε, Ιούνιο η Επίτροπος, η τον ομολογό της, Έγινε σε έργα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Τέλος πάντων πρόκειται για έναν τομέα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει και η αποστολή σας. Θα πάτε επίσης σε κάτι που έχει γνωρίσει προβολή, ε, δηλαδή κάποια αντιπλημμυρικά έργα ε, της πλημμύρας του 2014. Οπότε από εκεί φαίνεται το πόσο προσπαθεί η Ένωση Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, πληροφορίες και την ενημέρωση. θα τα αναζητήσουμε αυτά που μας είπατε, να τα δούμε όταν θα μεταβούμε επί τόπου. Τώρα εσείς παρακαλώ. Για τη Σερβία η κατάσταση είναι διαφορετική, ε, μάλλον για την Κροατία ε, η κατάσταση είναι διαφορετική από ό,τι εξήγησε η συνάδελφη για τη Σερβία. Η Κροατία είναι ήδη χώρα μέλος. Θα πω μία λεπτομέρεια σχετικά με την πολιτική κατάσταση εκεί, ότι πρόσφατα ε, σημειώθηκε κυβερνητική κρίση στην ε, Κροατία μετά από δύο πρόσφατες εκλογές. Με την, ε, σε αυτή την περίπτωση όμως επιλύθηκε η κρίση. Νομίζω εντάχθηκαν στην κυβέρνηση δύο νέοι υπουργοί και για την ώρα η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται. Εξετάζουμε βέβαια από τη δική μας σκοπιά την απορρόφηση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό που είναι σημαντικό για την Κροατία πρέπει να πω ότι η Κροατία πέρασε παρόμοιες καταστάσεις όπως μόλις περιγράφηκαν για τη Σερβία στην προενταξιακή περίοδο όμως από την 1η Ιουλίου 2013 όταν εντάχθηκε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, ε, άρχισε και η πρώτη περίοδος διαφθορτικών ταμείων για την Κροατία. Ε, περίοδος εκμαθήσεως κατά κάποιο τρόπο. Στην ουσία όμως, για να είναι κανείς ειλικρινής, περισσότερο μια παράταση της προεταξιακής περίοδου. Αλλά το 2014 είναι στην πραγματικότητα η πρώτη, ε, η έναξη μάλλον της περίοδου αυτής. Πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ορισμένα σημαντικά γεγονότα όταν αναλύει την κατάσταση, δηλαδή το γεγονός ότι η Κροατία λαμβάνει στην περίοδο αυτή τώρα το ενεαπλάσιο των ε, επιδοτήσεων. Εκεί χρειάστηκε να γίνουν πολύ σημαντικές προπαρασκευαστικές ενέργειες. Αυτές που ενδιαφέρουν περισσότερο είναι η στήριξη για τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας του συνόλου τη κρατική διοικήσεω και ιδίω σε ό,τι αφορά βέβαια την ε, διαχείριση ε, κοινοτικών κονδυλίων. Λαμβάνουν τώρα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ στην περίοδο αυτή, από τα οποία 6,8 τα διαχειρίζονται μέσα στα πλαίσια ευρυσιακών προγραμμάτων, η Γενική Διεύθυνση Regio είναι εδώ υπεύθυνη, ε, όπως γίνεται και στη Σερβία με σχετικά προγράμματα. Έχουμε και τη λεγόμενη κοινή διαχείριση, shared management, όπου ένα μέρος του management ανατίθεται στην, στις κρατικές αρχές και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με τις αρμόδιες αρχές επιτόπου, να σας παρουσιάσουν οι ίδιες οι αρχές τις πιο πρόσφατες δράσεις τους, αλλά και κάποια διορθωτικά μέτρα τα οποία λαμβάνουν με στόχο την βελτίωση της απορρόφησης και εφαρμογής των προγραμμάτων γιατί για να είμαστε ρεαλιστές όντως οι αριθμοί δεν ομιλούν υπέρ της Κροατίας δεν, είναι ε, απόλυτα ε, θετικοί ευνοϊκοί ορισμένα πράγματα όμως λαμβάνονται υπόψη όπως είπα ε, είναι το πιο, η πιο πρόσφατα ενταχθήσα χώρα μέλος και εκτός αυτού ένας αριθμός τομέων είναι απολύτως νέοι, διότι έως τώρα ήταν μόνο το περιβάλλον, οι μεταφορές, ανθρώπινοι πόροι και η γεωργία. Ενώ τώρα προστίθενται και άλλες προτεραιότητες για επενδύσεις, απολύτως νέες, απολύτως νέοι τομείς για τις αρχές που προωθούν τις κοινοτικές επενδύσεις, όπως για παράδειγμα ευρύ φάσμα, ε, δικαιονής ευρέως φάσματος, υγεία και ούτε καθεξής ε, παιδεία βεβαίω, που ήδη ενισχυόταν ε, κάτω από την οπτική των soft investment, αλλά τώρα βεβαίω είναι άλλα τα χρήματα. Τώρα, 74% της δημόσιας επένδυσης πηγαίνει στα πράγματα αυτά, πολύ σημαντικός αριθμός για να τον έχει κανείς υπόψη και δεν υπάρχουν τόσα θέματα εκεί σε ό,τι αφορά την ορατότητα των ευρωπαϊκών επενδύσεων όσο για τη Σερβία. Κάποια ερωτηματολόγια και κάποια δημοσκοπικά στοιχεία που διαθέτουμε δείχνουν ότι οι Κροάτες πολίτες αντιλαμβάνονται το μέγεθος των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Βέβαια δεν μας αρκεί η ε, κατάσταση αυτή και έτσι η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο συνεργάζεται με τις, ε, με τις κροατικές αρχές για να βελτιωθεί αυτή η εικόνα. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι η νομικοτεχνική και διοικητική βάση για την περίοδο αυτή, όχι μόνο για την Κροατία αλλά για όλες τις χώρες Υπάρχουν κάποια καινοτόμα στοιχεία σε σύγκριση με το παρελθόν. Πρόκειται για την εκ των προτέρων ερεσιμότητα, ex ante conditionality, που όροι πρέπει να πληρούνται ώστε μια χώρα μέλος να λαμβάνει πιστώσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα που συνήθως πρόκειται για μια στρατηγική βάση, δηλαδή εθνική στρατηγική σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, για να επωφεληθούν περισσότερο από τις επενδύσεις μας και να δοθούν προτεραιότητες που δεν δίνονταν πάντα. Και ο άλλο μηχανισμό τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης, είναι το πλαίσιο απόδοση performance framework. Εδώ υπάρχουν περισσότερες μετρήσεις ποιότητας, εισάγονται περισσότερες μετρήσεις ποιότητας, ώστε να είναι σε θέση μετά από κάποια περίοδο και στο τέλο τη περίοδου, δηλαδή τέλο 2018, και μετά τέλος 2023 να είναι σε θέση να μετρούν την ε, απόδοση, της ε, επιπτώσεις της πολιτικής συνοχής σύμφωνα με κάποιους δείκτες που θα πρέπει να ισχύουν ίδια για όλες τις χώρες μέλη, να μπορεί να μετρηθεί δηλαδή τι έχει επιτευχθεί έως τότε. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό λεπτομεριών θέλετε να προχωρήσω. Βλέπω όμως ότι θα συζητήσετε και με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι η Managing Authority η διαχειριστική αρχή δηλαδή για τα προγράμματα του, των διαφθορτικών ταμείων θα συζητήσετε και τα σχέδια δράσεως που είναι σημαντικά και οφείλω να πω ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στην Κροατία και μία από αυτές είναι ότι γίνονται τακτικά εκθέσεις από τη διαχειριστική αρχή προς την κυβέρνηση και μάλιστα ανά δύο εβδομάδες. Που τα θέματα αυτά εντάσσονται στην ατζέντα της κυβέρνησης. Δηλαδή έρονται σε υψηλό επίπεδο τα θέματα αυτά για να συζητηθούν. Και βλέπω επίσης ότι πρόκειται να επισκεφθείτε και έργα υποδομής που είναι και τα πιο ορατά ας πούμε έτσι για το κρατικό κοινό και τον απλό κρατη πολίτη. Επίσης όμως ένα καλό παράδειγμα είναι και το βιολογικό κέντρο. Κάτι που προσπαθούμε να προωθήσουμε ως μελλοντική επένδυση και όχι μόνο την πραγματική, την ειδική δηλαδή υποδομή, αλλά και επενδύσεις σε τεχνολογία, σε επιστημονική γνώση και είναι και ένα σημαντικό πράγμα που είναι η στρατηγική εφιούς ειδίκευσης. Αυτό καλούνται να το εφαρμόσουν όλες οι χώρες μέλη, ώστε να εξειδικευθούν και να δώσουν προτεραιότητα σε επενδύσεις, ιδίως στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας. Ευχαριστώ. Ωραία, ωραία, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ περιεκτικό. Ε, η Μαρτίνα. Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη ερώτηση. Έλαβα μόλις τώρα το ενημερωμένο πρόγραμμα και έκανα μια σύγκριση. Πρώτα ευχαριστώ τη Γραμματεία για το πολύ εξισορροπημένο πρόγραμμα, όπως πάντα. Νομίζω τα έχουμε εξισορροπήσει μεταξύ τους όλα. Να προσθέσουμε και κάποιες μη κρατικές οργανώσεις, τις οποίες δεν είδα, να τους επισκεφτούμε και αυτούς, διότι έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πανεπιστήμια, να βάλουμε και κάποιους μη, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό από τη δική μου πλευρά. Μήπως έρχεται και κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι πάντοτε χρήσιμο στις αποστολές αυτές να έχουμε και κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά νομίζω ότι ήδη περιλαμβάνεται όνομα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι καλό αυτό να είμαστε όλοι μαζί σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κάτι που θέλω να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Να αρχίσω με τη Σερβία, γιατί και εσείς αρχίσατε πρώτα με τη Σερβία. Θέλω να κατανοήσω καλύτερα ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να ρίξουμε περισσότερο βάρος και πού βρίσκονται πιο πολύ οι προκλήσεις. Είπατε ότι αναμένεται η επίσκεψή μας να βοηθήσει. Τι περιμένετε από την επίσκεψή μας, ποιος θα πρέπει να είναι ο πιο βασικός στόχος κάποιες προτάσεις. Επίσης επιθυμώ να ρωτήσω γνωρίζω ότι από τον τομέα των επιχειρήσεων. Αλλά θέλω να ρωτήσω τώρα και από την άποψη της, των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο διαδεδομένη είναι η διαφθορά. Ποια μέτρα λαμβάνονται κατά της διαφθοράς και τι άλλο μπορεί να γίνει. Τέλος, πώς εκτιμάτε την προστιθέμενη αξία των ε, ε, πόρων που διατέθηκαν στην προεταξιακή περίοδο. Και για την Κροατία, ίσως να λείπει ένα μέρος. Δηλαδή, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πράξη. Μιλήσατε για κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Τι κάνει στην καθημερινή βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπαιδεύει κόσμο, προσφέρει στήριξη, βοήθεια. Τα κάνει αυτά σε καθημερινή βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι είδους δείκτες εξετάζεται. Μιλήσατε για το ορόσημο του 2018. Αλλά τι μετρήσεις κάνετε τώρα. Τι είδους ε, δείκτες ελέγχετε. Και για την Κροατία, αν μου επιτρέπετε μια σημείωση προς την γραμματεία. Διότι θα γίνει ε, αποστολή και από την Επιτροπή Απασχόλησης στην Κροατία και πιο συγκεκριμένα για την, απασχόληση της, για την ε, πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων. Να μην βάλουν την Κροατία, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς ε, μπορεί να καλύψει την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Θα γίνει τον Σεπτέμβριο, εγώ όμως θα είμαι απούσα. Ε, σε μικρή ομάδα, γιατί πρόκειται για έκθεση ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να συντονιστούμε μαζί τους. Για να μην πηγαίνουν δύο αποστολέ από το Κοινοβούλιο για να συζητήσουν στην ουσία τα ίδια θέματα. Ας προσεγγίσουμε μια προσπάθεια συντονισμού. Ευχαριστώ. Α το εξετάσει η γραμματεία αυτό με τις μη κυβερνητικέ οργανώσει, αν μπορέσει να, να μπορέσουν να περιληφθούν. Τώρα, κάποιε κάποιες που έγιναν και από τη Μαρτίνα για την Σερβία. Μπορείτε να μας πείτε για την αποκέντρωση της διαχείρισης των κονδυλίων των ταμείων. Ήταν επιτυχής η προσπάθεια αυτή. Δεύτερο, αιρεσιμότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν ακυρωθεί κάποια έργα. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτά. Και να μας πείτε επίσης αν πρόκειται να συμμετάσχει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε και η Μαρτίνα, είναι χρήσιμο. Γιατί βεβαίω γνωρίζετε πολύ καλά τι χώρε αυτές και τα θέματα. Θα ήταν καλό αν κάποιος από την Επιτροπή μπορεί να μας συνοδεύσει. Ευχαριστώ. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να αρχίσω από την τελευταία. Η επιτόπου αντιπροσωπεία μας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο και θα σας ε, συνοδεύουν σε όλο το ταξίδι σας. Η δε επιλογή των έργων που θα επισκεφτείτε έχουν, έχει γίνει σε συνεργασία μαζί τους. Θα είναι μαζί σας και θα σας δίνουν ό,τι πληροφορίες χρειαστείτε. Για τις ε, μείζονες προκλήσεις για την Σερβία και την απορρόφηση των πόρων. Η πρόκληση αρχικά ήταν ότι θα κάνουν τα πράγματα αυτά για πρώτη φορά. Όταν άρχισε η εφαρμογή το 2013 ήταν κάτι απολύτως νέο για αυτούς και μέγα ποσοστό του προγράμματος δόθηκε για άμεση διαχείριση του έργους. Ήταν λοιπόν σημαντική πρόκληση. Από τότε η πρόκληση είναι η εκπαίδευση και η διατήρηση του προσωπικού. Για όλη τη διοίκηση δεν ισχύει αυτό. Όχι μόνο για ευρωπαϊκές δομές, πρόκειται για οριζόντιο πρόβλημα το οποίο το αντιλαμβανόμαστε και το βλέπουμε ιδίως από τη δική μας πλευρά, σε ό,τι αφορά την ε, ένταξη, την προοπτική ένταξη δηλαδή. Όμως είναι κάτι που διατρέχει την ε, διοίκηση, είτε πρόκειται για προσωπικό το οποίο αναμειγνύεται σε ζητήματα ευρωπαϊκά είτε όχι. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν κάποιες προτεραιότητες ε, για λειτουργίες που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση συντονισμό μεταξύ των πολιτικών στόχων της, Ευρωπαϊ... της, ε, της Σερβίας και τον αριθμό ανθρώπινων πόρων που ε, δίνονται. Όταν λέω ότι θα βοηθήσει η αποστολή σας, το λέγω διότι θα τονίσει τη σημασία που αποδίδουμε για ε, την απόδοση της στήριξης που δίνουμε στη Σερβία και βεβαίω και την ορατότητα της στήριξης που δίνουμε. Θα ασχολείται ιδίω με το πώς δαπανούν τα χρήματα που τους διαθέτουμε και την προτεραιότητα που δίνουν σε στήριξη για την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα κράτους δικαίου, δημόσιας διοίκησης. Το μήνυμα αυτό είναι σημαντικό να περάσει στους Σέρβους πολίτες για την διαφθορά αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Σερβία. Αναφέρθηκα σύντομα στο monitoring που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το κράτος δικαίου γενικότερα και ένας από τους τομείς όπου και εμείς και οι χώρες μέλη συζητούμε και διαπιστώνουμε ότι πρόκειται εκεί πράγματι για μείζωνα πρόκληση η διαφθορά. Υπάρχει συμβούλιο κατά της διαφθοράς, υπάρχει νέα νομοθεσία κατά της διαφθοράς που έχει εγκριθεί αλλά που κάπου έχει κολλήσει μέσα στο σύστημα. Πρόκειται λοιπόν για πρόοδο η οποία οφείλει να γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τομέα αυτό. Για το ερώτημα σε ό,τι αφορά την μέτρηση της προστιθέμενης αξίας. Ότι όντως αυτά που κάνουμε δηλαδή αποδίδουν επιτόπου στην προσπάθεια ένταξης, πορείας προς την ένταξη. Μετρούμε δηλαδή την απόδοση σχετικά με τους καθαρούς στόχους και δείκτες ΕΙΠΑ δύο και στο επίπεδο των δράσεων. Εκεί υπάρχουν καθαροί δείκτες και δράσεις. Θέλουμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι μπορούμε να επιτύχουμε και να το παρακολουθούμε καθώς αναπτύσσονται τα προγράμματα και τα έργα. Αυτό είναι το πλαίσιο απόδοσης και τα baselines. Και τέλος η ανταμοιβή απόδοσης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά όπου ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να αποδώσει την απόδοση, να αντικατοπτρίσει δηλαδή την απόδοση ολόκληρης της χώρας. Εκεί εσείς κύριε Πρόεδρε ρωτήσατε, αν η αποκεντρωμένη διαχείριση αποτελεί επιτυχία. Ακόμα είναι νωρίς να το πει κανείς αυτό ακόμη. Το πρώτο ε, πρόγραμμα άρχισε το 2013 και ακόμα δεν έχουμε καν ολοκληρώσει τις αναθέσεις. Έχουμε και πολύ λίγο προσωπικό που συνεργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Τους τελευταίους μήνες και χρόνια όμως έχουν αφιερώσει περισσότερους πόρους από πλευρά Σερβικής και οι συζητήσεις που διεξάγουμε μαζί τους και εδώ στις Βρυξέλλες αλλά και επί τόπου. Ε, νομίζω τώρα έχουν αναπτύξει καλή ικανότητα που πρέπει όμως να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα, πολύ σημαντικό θέμα. Το συνδέω και πάλι με την ορίμανση των έργων. Έχουμε διδαχθεί από την εμπειρία ότι όπου υπάρχουν υπερβολικά πολλοί όροι αιρεσιμότητες στην αρχή των έργων που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πληρωθούν οι όροι αυτοί και επομένως να μην επιτυχές το έργο. Βάζουμε τώρα για κάποιους σε μια πιο ύστερη περίοδο, ώστε να υπάρχει λιγότερο κίνδυνο ε, να αποτύχουν στην πλήρωση ορισμένων όρων. Για την ώρα φαίνεται πάντω αυτή η προσπάθεια να κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Για την Κροατία τώρα, τι μπορείτε να μα πείτε. Ε, πρώτη σα ερώτηση σχετικά με το τι κάνει σε καθημερινή βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει την διοικητική ικανότητα. Μπορώ να σα αναφέρω βεβαίω όχι εξαρτητικά διάφορε δράσει πέραν των άμεσων διασυνδέσεων και της άμεσης ενίσχυσης πραγματικά μέρα με την ημέρα από την κάθε γεωγραφική μας μονάδα προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Στη DG Regio υπάρχει και μια οριζόντια μονάδα η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την διοικητική ικανότητα της ε, Κροατίας και αναπτύσσουν διάφορα έργα, εργαλεία συγγνώμη, για να βοηθήσουν όλες τις χώρες μέλη οι οποίες έχουν ανάγκη. Βάσεις δεδομένων ε, δεξιοτήτων, με περιγραφές ε, καθηκόντων για τις διάφορες θέσεις, για όλα τα αναγκαία προφίλ θέσεων, για τις αρχές οι οποίες ε, παρακολουθούν τις επενδύσεις. Το δεύτερο είναι η αξιολόγηση ομοτήμων, peer-to-peer. -peer. Συνήθως αυτό δεν ε, περιλαμβάνει δημοσιονομική βοήθεια, αλλά ανταλλαγή εμπειριών. Ανταλλαγή εμπειριών ε, μεταξύ χωρών μελών που τα καταφέρνουν καλά σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, ε, να συνεργαστούν δηλαδή σε, με χώρε μέλη που έχουν ανάγκη σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Εξάλλου, σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα υπάρχει χώρος για τεχνική συνδρομή που περιλαμβάνει σαφώς περιγραφόμενα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, βεβαίως και εκπαίδευση του προσωπικού, όπως είπατε και εσείς. Παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις δράσεις που, στις οποίες προβαίνει η διαχειριστική αρχή. Το καλό νέο για την Κροατία είναι ότι τον Μάιο ελήφθη απόφαση από την κυβέρνηση να διαθέσει, μάλλον να προσλάβει 600-650 ανθρώπους σε τομείς οι οποίοι εμπλέκονται σε ζητήματα ε, διαφορετικών ταμείων. Επίσης ζητήματα θαλάσσιας οικονομίας, αλληλεία, γεωργία Βέβαια η πρόσληψη απλώ προσωπικού δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά έγινε ένα βήμα. Και επιτρέπει σε κάποιες διαδικασίες να γίνονται πιο απλές, συντομότερες, αφού βέβαια η πρόσληψη ε, προσωπικού δημοσίων υπαλλήλων δηλαδή είναι χρονοβόρα. Προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα αυτό όσο γίνεται πιο απλά, βεβαίω τηρώντα τον νόμο. Δεν υπάρχει εμβολία άλλα άλλη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι για παράδειγμα σε συγκεκριμένα θέματα όπως κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες προμήθειες όπου εκεί υπάρχουν, υπάρχει ε, οριζόντια, ε, οριζόντια αιρεσιμότητα για, την, για τις ε, δαπάνες ευρωπαϊκών κονδυλίων με σχέδια δράσεως που αναπτύσσει η κυβέρνηση που περιλαμβάνουν εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων που εμπλέκονται στην ε, χρήση των κονδυλίων που διαθέτουν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Και σε ό,τι αφορά ε, τα μέτρα υποδομών, η DG Regio συνεργάζεται στενά αλλά και πληρώνει προσωπικό, ομάδες, του συστήματος Jaspers και που ενισχύουν την προσπάθεια των κρατικών αρχών. Επίσης, γίνονται και παρεμβάσεις SRSP που είναι το νέο όργανο της Κομισιόν που χρηματοδοτεί επίσης και εφαρμόζει ορισμένα έργα αν και δεν έχει δοθεί ακόμη τελική μορφή εξ όσων γνωρίζω θα γίνουν κάποιες ενδοϊπηρεσιακές διαβουλεύσεις την επόμενη εβδομάδα πάντως σε κάποια έργα τα οποία αναφέρονται επίσης στην διοικητική ικανότητα για την πρώτη σας ερώτηση. Για Δεύτερη, ίσως έδωσα κάπως επιφανειακή εικόνα του τι κάνουμε για να αξιολογήσουμε την πρόοδο της εφαρμογής. Δεν μιλούμε μόνο για το 2018 έως 2023. Εκεί είναι πάντως οι πιο γενικές αξιολογήσεις που θα γίνουν μέσα στο πλαίσιο του δικτύου απόδοσης. Για την Κροατία πιο συγκεκριμένα γίνονται τριμηνίες εκθέσεις, υποβάλλονται τριμηνίες εκθέσεις, εκθέσεις που στέλνουν οι αρχές στην κυβέρνηση, διάφορες αρχές στην κεντρική κυβέρνηση, πρόκειται για, πρώτα για εσωτερικές εκθέσεις, αλλά έρχονται και σε εμά. <coughs> και στο τέλος της εβδομάδας ή στο τέλος του μηνός θα έχουμε και ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής για το πρόγραμμα που θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε την πρόοδο. Αυτά είναι αριθμιστικά μέτρα, αλλά είμαστε πραγματικά καθημερινά σε επαφή με τις κρατικές αρχές διεξάγουμε κοινέ τεχνικέ συναντήσει και παρακολουθούμε πολύ στενά την πρόοδο. Σα ε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα είδατε στο σχετικό σήμερα διάταξη στο πρόγραμμα, αλλά θα υπάρξουν και κάποιε μικροδιορθώσει ανάλογα δηλαδή με τα όσα θα αποφασίσουμε και ευχαριστούμε τη γραμματεία ε, που σύνταξε αυτό το πρόγραμμα και ευχαριστούμε και την Επιτροπή μας ε, έδωσε περαιτέρω διευκρίνησης. Άρα λοιπόν τώρα περνάμε στο σημείο που αφορά την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την, ε, την Ισία. Ο κύριος ε, Πίνξτεν λοιπόν να πάρει το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεση του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε members of this committee. Ξέρουμε λοιπόν μέλη της ε, Επιτροπής, θα θυμόσαστε όλοι ότι τον Ιανουάριο του 2011 είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο της ε, Αραβικής Άνοιξης η Evolution, Jasmine Revolution. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δεσμεύσει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ε, για την περίοδο 2011 έως 2015 για την, ε, την Ισία με δύο στόχους. Να διευκολύνει τη δημοκρατική μετάβαση ε, και δεύτερον να υποστηρίξει την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτοί λοιπόν, αυτοί ήταν οι δύο κύριοι στόχοι της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την, τον έλεγχό μας ε, ακολουθώντα μια δομή τεσσάρων θεμάτων, δηλαδή κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την ίδια την έκθεση, μετά παρατηρήσεις, τι διαπιστώσαμε, μερικά πράγματα σε ό,τι αφορά το ΕΦΑ και από εκεί και μετά συμπεράσματα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με το τι περιλάμβανε αυτή, αυτός ο έλεγχος. Κατά πόσο δαπανήθηκαν σωστά, αν θέλετε, τα εν λόγω κονδύλια. Αυτός ήταν ο στόχος, δηλαδή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του, των, των, κονδυλίων που κατευθύνθηκαν προς την Τινησία. Και εδώ δηλαδή εξετάσαμε κατά πόσο ε, η Επιτροπή ανταποκρίθηκε σωστά στις κύριες προκλήσεις που αντιμετώπιζε την Ισία και δεύτερο υπό ερώτημα αν θέλετε ε, ήταν το κατά πόσο η εκτέλεση εδώ των σχετικών προγραμμάτων ήταν σωστή ή όχι. Να σας πω επίσης ότι το δείγμα ε, του ελέγχου ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο αφού κάλυψε το 70% του συνόλου της ε, υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισία. Τι ελέγξαμε εδώ. Ε, ε, ελέγξαμε το δάνειο MFA, δηλαδή μακροοικονομική υποστήριξη, 300 δις ευρώ και τέσσερα προγράμματα υποστήριξης προϋπολογισμού και ε, αναλύσαμε και 14 project έργα. Αυτά λοιπόν ως προς το τι περιείχε αυτή η, αυτός ο έλεγχος, αυτή η αξιολόγηση. Τώρα, Ποια είναι τα πορίσματα, τι βρήκαμε. Θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και η Επιτροπή πράγματι ασχολήθηκαν ή αν θέλετε κατεύθυναν τα κονδύλια ε, προ τι κύριε προκλήσει που αντιμετωπίζει την ΕΣΕ. Επίση, τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν σημαντικά, όπω θα ανέμενε κανεί, μέσω πέντε γενικών προγραμμάτων υποστήριξη του προπολογισμού Ε, των ΠΑΣ όπως λέγονται. Εδώ είχαμε να κάνουμε με λίγο παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ και από εκεί και μετά ε, είχαν εξαπλωθεί αν θέλετε σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό ε, πεδίων ε, ή θεματικών ε, πεδίων το, τα εν λόγω κονδύλια. Αν δείτε δηλαδή τη σχετική έκθεση θα διαπιστώσετε ότι είχαμε 20 τομείς οι οποίοι αναφέρονται. Και υπήρχε παρόλα αυτά γενική συνένεση ότι τουλάχιστον ή μάλλον το, κατά το μέγιστο τρεις ε, τομείς είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να υποστηριχθούν. Οπότε δεν ήταν αρκούντος στοχευμένη η προσέγγιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συντονισμό με τους ε, χορηγούς, άλλους χορηγούς, δηλαδή την ε, Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και ούτω καθεξή, ήταν καλός εδώ ο συντονισμός με τους υπόλοιπου χορηγού, αλλά από την άλλη εάν δείτε την, τον κοινό προγραμματισμό με τα κράτη-μέλη, εδώ δεν υπήρξε καλό συντονισμό παρότι δηλαδή προβλέπεται στον κανονισμό ΕΝΑΡ, δεν υπήρξε κοινό προγραμματισμό με τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, την γενική δημοσιονομική υποστήριξη του προπολογισμού, να πούμε ότι εκταμιεύθηκε ταχαίω, όμω σε έναν υπερβολικά ευέλικτο, με έναν υπερβολικά ευέλικτο τρόπο. Ω προ δηλαδή τι ε, προποθέσει οι οποίε έπρεπε να πληρούνται, διαπιστώσαμε ότι ενίοτε οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονταν στις συμφωνίες χρηματοδότησης ήδη πληρούνταν κατά την χρονική στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας ή, εν πάση περιπτώσει, οι αξιώσεις ή οι προϋποθέσεις ήταν πολύ ε, μετριασμένες, αν θέλετε, και ήταν πολύ εύκολο δηλαδή να τα αποκλειστεί σε αυτές η την Για παράδειγμα, εάν θέλει κανείς να παράσχει κάποια κίνητρα σε μια κυβέρνηση, τότε δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά μαλακός, υπερβολικά ευέλικτος ως προς τις προϋποθέσεις ε, που θέτει στο επίπεδο της διακυβέρνηση. Εάν δηλαδή ε, αναμένει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, ε, στις οποίες θα πρέπει να προβεί η ενδιαφερόμενη ε, κυβέρνηση, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, δημόσια διαχείριση ή την καταπολέμηση της διαφοράς ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να παρέχει κανεί τα κατάλληλα κίνητρα, ούτως ώστε οι προϋποθέσεις να μην είναι πολύ μετριασμένες. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τις αιρεσιμότητε στο πλαίσιο της υποστήριξης του προπολογισμού. Από εκεί και μετά η αξιολόγηση του είναι πάρα πολύ σημαντική και όπως μπορεί κανείς ε, να διαπιστώσει διαβάζοντας την έκθεση, τα πορίσματα σε ό,τι αφορά την τελευταία αξιολόγηση των ΠΕΦΑ, σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθυνών, σε ό,τι αφορά την ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, θα διαπιστώσουμε ότι μόλις δηλαδή εκταμιευθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια και φτάσουν σε αυτό το επωνομαζόμενο black box, ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πράγματι έχουν ταπανηθεί με τον κατάλληλο τρόπο αυτά τα κονδύλια. Δηλαδή, είχαμε μία τέτοια ε, πέφα το 2010 και μετά μία το 2015 και μετά μια φέτος η οποία όμως αφορούσε μόνο την περίοδο 2011 έως 2013 που βέβαια είναι πολύ παλιά οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση πέφα. Από εκεί και μετά αυτό που ανέφερε η Επιτροπή ως απάντηση στη σελίδα 56 σε ό,τι αφορά το ΠΕΦΑ και όπου λέει δηλαδή δεν εξαρτάται από την Επιτροπή ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό εξαρτάται από την επιχείρηση εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση από την κυβέρνηση της Τινεσίας να πω ότι ναι μεν αυτό ισχύει μέχρι ενός βαθμού αλλά για να είμαι ταυτόχρονα και πολύ ειλικρινής μαζί σας είναι πολύ ε, όλο αυτό το επιχείρημα δηλαδή η αξιολόγηση ΠΕΦΑ, είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να την εξετάσει προσεκτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προφανώ από κοινού την Επιτροπή. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση ΠΕΦΑ, τόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση τη νησία, όσο και γενικότερα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ε, αξιολόγηση ΠΕΦΑ όπως αυτή διεξήχθη ή τελικά δεν διεξήχθη στην περίπτωση της ε, όπως διεξήχθη, εν πάση περιπτώσει, Τώρα, κλείνοντας, Πρόεδρε, ποια είναι τα συμπεράσματα αυτού του ελέγχου. Και εδώ θα επαναλάβω κάποια από τα στοιχεία που ήδη ανέφερα, μόνο και μόνο για να υπογραμμίσω τη σημασία τους. Θετικά, λοιπόν, ε, συμπεράσματα, γενικά δαπανήθηκαν με το σωστό τόπο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τινησία. Τα ε, κονδύλια λοιπόν συνέβαλαν σημαντικά στους δύο, στην εκπλήρωση των δύο κυρίων στόχων, δηλαδή μετάβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα και οικονομική σταθερότητα. Αυτό λοιπόν επιτεύχθηκε και εγκαίρως μάλιστα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η Επίτροπη, η προσέγγιση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ήταν πολύ φιλόδοξη και καλό είναι να είναι καλή σε φιλόδοξε, αλλά υπερβολικά μεγάλο αριθμών προτεραιοτήτων καλύφθηκε και όπω ήδη είπα δεν ήταν αρκούντο στοχευμένη η επένδυση των κοντιλίων. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τον συντονισμό με του άλλου χορηγού, ναι, έγινε πολύ καλά και μπράβο στην Επιτροπή, αλλά από την άλλη πλευρά ο κοινό προγραμματισμό με τα κράτη-μέλη, όπω προβλέπεται και στον κανονισμό, δεν ήταν ικανοποιητικό. Οπότε εδώ θα πρέπει να γίνουν βελτιώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα προγράμματα υποστήριξη του προπολογισμού και δεν περιείχαν και συνεχίζουν να μην περιέχουν τα κατάλληλα κίνητρα απέναντι στις αρχές ε, της θυνησίας. Όπως σας είπα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι προϋποθέσεις ήδη πληρούνταν όταν δηλαδή υπογράφονταν η σχετική συμφωνία. Ή σε άλλες περιπτώσεις οι εν λόγω προϋποθέσεις ήταν υπερβολικά ευέλικτες. Όπως συμβαίνει, θα πρέπει να πω, γενικά. Όχι δηλαδή σε σχέση με αυτή τη χώρα, αλλά και σε πολλούς άλλους ε, ελέγχους όταν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ε, ε, υποστήριξη του προπολογισμού. Ακόμα λοιπόν και στις περιπτώσεις όπου οι προϋποθέσεις δεν πληρούνταν ή ήταν υπερβολικά ευέλικτες, παρόλα αυτά οι εκταμιεύσεις των κονδυλίων γίνονταν. Οπότε, λαμβάνοντα υπόψη την υψηλή υποστήριξη του προπολογισμού που υπερεύει το μισό δις από το 2010 και καθώς τότε δεν υπήρχε και αξιολόγηση ΠΕΦΑ, θα πρέπει να πούμε πως το συμπέρασμά μας δεν ικανοποιητική κατάσταση για να μην πω είναι απολύτως ε, απαράδεκτη. Τώρα σε ό,τι αφορά το ε, δάνειο των 200 εκατομμυρίων ευρώ MFA, δηλαδή της μακροοικονομικής ενίσχυσης, να πούμε πως ε, πραγματικά ήταν απολύτως απαραίτητη η εν λόγω υποστήριξη και εκτάκτως απαραίτητη. Παρόλα αυτά όμως, ότι διαπιστώσαμε ότι ε, χρειάστηκαν δύο χρόνια τελικά για να ε, διατεθεί. Και βέβαια θα μπορούσε κανεί να πει ότι είναι, αυτό οφείλεται στην Τινησία, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάστηκαν 11 μήνε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να χορηγηθεί αυτή η υποστήριξη και είναι υπερβολικά μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και επιτρέψτε μου τώρα, ε, Πρόεδρε, να σχολιάσω λίγο και το σχετικό έγγραφο του ε, συγκητή σας. Ε, δηλαδή πραγματικά ε, συγχαίρω τον συγκητή σας τον κύριο Παρνιό. Πραγματικά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Και θα πρέπει να συγχαρώ και τα μέλη σας. Για το συμπέρασμα, για τις συστάσεις τις οποίες συμμερίζομαι 100% μπράβο, μπράβο για τον έγγραφο σας επί των τύπων των ύλων. Εφέσατε τον δάκτυλο. Ακριβώς ως αυτά τα οποία λέτε αντιστοιχούν 100% είναι αυτά που ξέρουμε κι εμείς. οπότε, ξέρετε, εγώ διάβασα το κείμενό σας αφού εγώ διαμορφώσα κάποια άποψη. Οπότε νομίζω ότι η δουλειά σας είναι πολύ ψηλό επίπεδο και συμφωνούμε με συστάσεις και με συμπεράσματα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Αυτά για σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε ως συνήθως πάρα πολύ ολοκληρωμένη παρουσιασή σας. Συγχαρητήρια. Α, ως συνήθως είπατε. Μπράβο, μπράβο. Και ο κύριος Παρνιό έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Επίσης τον κύριο Καρέλ, από το Ελληνικό Συνέδριο που πάρα πολύ ευχάριστα τα, είπατε και ναι, όντως έχουμε αυτές τις συστάσεις με τις οποίες συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι οι ευρωβουλευτές, όλοι όσοι θελήσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την ε, προσπάθεια ε, και οι ισχυώδεις εισηγητές που θα λάβουν στη συνέχεια τον λογό ο κύριος Τομάς από το ΕΛΚ. Μας είπατε για το πόσο είναι σημαντικό να αναδείξουμε ε, το ότι είναι πολύ πλήρης η εκθεσή σας και εγώ με τη σειρά μου συμφωνώ με συστάσεις και συμπεράσματά σας. Άκουσα την εισήγησή σας αφού είχα συντάξει τη δική μου έκθεση και η ομοιότητα είναι μεγάλη όσον αφορά την προσέγγιση μας και έχω εντάχει να σας πω για κάποια σημεία όπως είπατε και εσείς σημαντικό να τονίσουμε ότι έχουμε αυτά τα τρία δις τα οποία εγκρίθηκαν για την, ε, την νησία και τα οποία έπιασαν τόπο. Ε, όπως τα είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πενθυμίζουμε και να πούμε επίσης ότι τα ευρωπαϊκοί πόροι βοήθησαν στον δημοκρατικό μετασχετισμό για τη χώρα, για τη σταθεροποίηση της οικονομίας μετά από την επανάσταση του Γιασεμνιού του 2011. Πολύ σημαντικό και αυτό να το υπενθυμίσουμε. Επίσης έχουμε τις πολιτικές συστάσεις του εγγράφου εργασίας που σας παρουσιάζω από πλευράς της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και λέμε ότι πάρα πολύ σωστός ήταν ο συντονισμός μεταξύ των ε, χρηματοδοτών του ε, νομισματικού ταμείου, της Παγκοσμίου Τράπεζας, τέλος πάντων της Τράπεζας Επενδύσεων, της ΕΤΕ και ε, όπως είπε και το ελεγκτικό συνέδριο ιδιαίτερα η Γαλλία και η Γερμανία βελτίωσαν τον συντονισμό όσον αφορά τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο τις αρχές της χώρας. Αλλά πρέπει να εστιαστεί η Ευρώπη σε λιγότερους στόχους, σε λιγότερους τομείς, αλλά να τους περιχαρακώσει, να τους ξεκαθαρίσει περισσότερο και έτσι επομένως αυτή η τομιακή βοήθεια θα βελτιωθεί εάν ε, οι προτεραιότητες ξεκαθαριστούν, αλλά να ξεκαθαριστούν και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις Επομένως έχουμε μια πιο καλά διαρθρωμένη, στοχευμένη πρωτοβουλία από την Ευρώπη. Για όλε αυτέ τι μεταρρυθμίσει που τώρα ζητηθεί η δικασία ολοκλήρωση, πάντω θα πρέπει να πούμε και κάτι συγκεκριμένο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πούμε ότι στην έκθεση του το, Ευρωπαϊ... το Ελληνικό Συνέδριο ε, λέει ότι δυστυχώ είχαμε την τελευταία αξιολόγηση. Μα τίποτα στην προσωπική εισήγηση. Ότι λέτε για τι ε, δαπάνε, για το ΠΕΦΑ που ανάγεται στο 2010 και κατά τη γνώμη μα. κατά τη γνώμη σα αυτό είναι το καλύτερο μέσο τόσο ώστε να αξιολογήσουμε το πώ έχουν προχωρήσει οι μεταρρυθμίσει και τα δημοσιονομικά και βέβαια όπω είπατε ε, είχαμε ε, την αξιολόγηση του 2014 που αναβλήθηκε για τον Μάρτιο του 2017 οπότε πέστε μα από πλευρά τη Επιτροπή, τι έγινε με αυτή την αξιολόγηση τι δημοσιοποιήσατε μα αν είναι έτσι, να μας πείτε σε τι συμπεράσματα καταλήξατε. Αυτά έχω να πω. Συνάδελφοι, ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παρνία. Ο κύριος Τόμας. Κύριος Σντεχόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, θεώρησα ότι μπορώ να σας τα πω τσέχικα. Είπατε Τέλος, με το μικρό το μόνο που με φανάξατε, σας ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο. Πάρα πολύ κατανοητό το κείμενο και έχει πολλά στοιχεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε στο μέλλον για τις αξιολογήσεις μας. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κύριο Παρνιό και το έργο είναι αξιόλογο και η έκθεσή του. Νομίζω ότι ξέρει τα θέματα καλά και επίσης θέλω να σταθώ στα εξή σημεία. Έχουμε αυτή την αρρωγή προς τις γενικέ χώρες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως όσον αφορά την πτυχή ασφάλεια. Η τίνηση είναι πολύ σημαντικό σε και όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά και για τα θέματα ασφαλείας. Οπότε, και είναι πολύ σημαντική βοήθεια που χορηγούμε εμείς στην χώρα. Βασική προτεραιότητα είναι να υπάρχει μακροπρόθεσμα σταθερότητα, ε, χρηστή διοίκηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη χώρα. Και αυτό θα επηρεάσει όλη την περιοχή αλλά και τις μακροπρόθεσμες σχέσεις μας. Είναι επομένως ακόμα πιο σημαντικό να υπάρχει συνεργασία και έτσι να λύσουμε τα προβλήματα της ασφαλείας, τα προβλήματα για τη μετανάστευση, ε, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και να μπορέσουμε να διαλύσουμε τα δίκτυα των τρομοκρατών. Είπαμε ότι περνάει έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό τώρα η χώρα και όπως και στο Μαρόκο μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών έχουν περάσει από αυτή την διαδρομή οπότε μπορούμε να εισφέρουμε τη δική μας ε, εμπειρία, τη δική μας γνώση στη χώρα. Δυστυχώς ακόμα παλεύει με προβλήματα η νησία. Αυτό δεν διευκολύνει το έργο της ε, χώρας. Δηλαδή έχουμε ανισότητες οικονομικές και κοινωνικές, έχουμε ανεργία κυρίως για τους νέους, έχουμε και περιθωριοποίηση στην Τινησιακή κοινωνία. Για όλα αυτά μπορούμε να βοηθήσουμε. Τέλος πάντων, για να ξαναγυρίσουμε τα θέματα του οικονομικού ελέγχου, σωστά λέει το Ελληνικό Συνέδριο ότι οι ευρωπαϊκοί υπόροι πιάσαν τόπο στην ε, ε, την Ισία και πάρα κάποια προβληματάκια αξιοποιήθηκαν την επόμενη φορά. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα καθορίσουμε και τις προτεραιότητες και να μην πάνε πόρε σε πάρα πολλές υπερβολικά πολλούς τομείς. Καλύτερα να επικεντρωθούμε σε λιγότερους στόχους, λιγότερους τομείς και εκεί να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει περισσότερο τα χρήματα, να βρει την ε, σταθερότητα και έτσι να μην έχουμε λιγότερα χρήματα αλλά σε περισσότερους τομείς. Αυτό το να το συναντούμε σε πολλές χώρες που βοηθά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τη ρόλο θα αναλάβει να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε, χαρακτήρα επιδότησης των ε, ενισχύσεων μας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και πλάσεις ανθρωπίνων πόλων την χώρα. Έχουν υπάρξει επικρίσεις στο παρελθόν ότι κάνουμε λίγα. Δεν βοηθούμε με την εμπειρία μας ε, τη χώρα, για παράδειγμα, κατά της διαφοράς, κατά του οργανωμένου κλίματος, για ας να βοηθήσουμε διάφορες περιφέρειες να αντιμετωπίσουν την εξηρασία και είναι πολύ η την που μεταναστεύουν, μετακινούνται μάλλον γιατί δεν έχουν πόσιμο νερό. Έχουμε το Erasmus Plus και αυτό είναι προτεραιότητα σε σχέση με το Horizon 2020. Πρόκειται για προγράμματα που έχουν ριζώσει στη χώρα πολύ καιρό, μεγάλη ήταν η επιτυχία τους, όμως είναι σημαντικό ζήτημα η ασφάλεια και η τρομοκρατία. Αυτά τα προβλήματα χτυπάνε και τον τουρισμό και την οικονομία της χώρας. Οπωσδήποτε πρέπει να τύχουν προτεραιότητες. Και προς τα εκεί θα πρέπει να πάει η ευρωπαϊκή βοήθεια. Να υπάρχει επίσης ευελιξία. Νομίζω ότι η χώρα τα πάει καλά όσον αφορά την προστασία των συνόρων, όσον αφορά τον έλεγχο της μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Βοηθά τις επιχειρήσεις διάσωσης. βοηθά για διάφορα θέματα των υπηρεσιών πληροφοριών, στρατηγικούς τομείς. Για να μην ξεχνούμε και την κοινωνία των πολιτών. Έχει βοηθήσει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια εκδημοκρατισμού της χώρας. Ταχαίως πρέπει στην Τινησία να προχωρήσουμε με μέτρα για τη μετανάστευση κατά της τρομοκρατίας γιατί δεν έχουν προχωρήσει με τόσο γρήγορους ρυθμού στο παρελθόν παρά το ότι η έγκριση αυτών των μέτρων έλαβε χώρα ταχαίως. Κλείνοντας να σας πω ότι πιστεύω πως η έκθεση θα βοηθήσει. Ούτως ώστε οι χώρες της Βορειοαφρικής να αξιοποιήσουν την ε, ενίσχυση από πλευράς μας. Θα πρέπει να είναι όμως στοχευμένη. Θέλουν τις χώρες να συνεχιστεί η συνεργασία. Δεν χρειάζεται χωρί ξεχωριστή πολιτική, δεν χρειάζεται να αναζητήσουν βοήθεια χτύποντας την πόρτα της Ρωσίας. Γιατί οι υποσχέσεις είναι ε, φρούδες από εκεί. Ευχαριστούμε. Τόμας, λέει ο πρόεδρος. Δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά στα τσέχικα. Ε, ίσως μπορώ να πω λίγες λέξεις μόνο, αλλά αυτό είναι όλο. Η Μαρτίνα. Εγώ θα μιλήσω τώρα εξ ονόματος του Χάνου Τάκουλα που είναι ο σκιώδης μας του, των φιλελευθέρων και μου έχει πει να σας πω τα εξής ε, ερεσιμότητα σημαντική κριτήριο για τη χρηματοδότηση άλλων χωρών θα πρέπει να είναι σαφές το μήνυμα αυτό όπως στην περίπτωση της Ενησίας όπου βλέπουμε για παράδειγμα προγράμματα PAR που χρησιμοποιούνται, που ε, χρηματοδοτούνται για χρόνια. Θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά οι εξελίξεις. Έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητούμε πρόοδο ως προϋπόθεση, ως όρο για την περαιτέρω χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε αξιολόγηση των προγραμμάτων για να μην δίνεται εντύπωση ότι δεν παρακολουθείται η εφαρμογή ε, των προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα αυτόματο ταμείο όπου καθένας προσέρχεται και λαμβάνει χρήματα. Καλύπτονται διάφοροι τομεί. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνολική αξιολόγηση της συνεργασίας. Και ο δε μα ευχαριστεί και το ελεγκτικό συνέδριο τον κύριο Πίνξτεν και τον εισηγητή κύριο Πανιού για το έργο τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλλερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω είναι παρόν και ας ακούσουμε τι έχετε να πείτε και ιδίως απαντήσει τις ερωτήσεις που έχουν θέσει οι βουλευτές μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εσάς κύριε Σιγητά και εσάς κύριε Πίνξτεν. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευχαριστώ απόγευμα διότι πρόκειται για μια από τις ε, πιο ε, μια, ε, τις καλύτερες που έχω δει από το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και βεβαίω και η έκθεση του Πάνιο. Ο Πίνξτεν είπε πριν λίγο ότι παρά την κριτική που ασκεί για ορισμένε λεπτομέρειες, ότι τα χρήματα αυτά έχουν δαπανηθεί σωστά. Η έκθεση είναι θετική στο σύνολό τη. Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση που κάνει είναι πολύ επικοδομητική και ευχαριστώ με την ευκαιρία τον κύριο Πίνξτεν και την ομάδα του για την θαυμάσια συνεργασία που είχαμε ε, και για την εσύνταξη εκθέσεως, η οποία έκθεση λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρά ταχαίως και αποτελεσματικά στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή, η Τινησία δηλαδή, στην πρόσφατη περίοδο. Και είναι σαφές νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές που έχουν διέλθει από παρόμοιες εμπειρίες στις χώρες τους, όπως ο κ. Στεχόσκι, που είναι Τσέχος και έχει περάσει και η χώρα του τέτοιες ταραχώδεις ε, περιόδους, αυτή η μετεπαναστατική περίοδος που ζει η Τινησία είναι μια ε, περίοδος γεμάτη προκλήσεις. Μεταξύ αυτών και οικονομικές και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων. Για φανταστείτε μια χώρα όπου μέσα σε έξι χρόνια πέρασε 7 διαφορετικές κυβερνήσεις. Με σε μια τέτοια κατάσταση δεν είναι και προφανές ε, να βάλει κανείς προτεραιότητες, να επιβάλλει όρους για την χρήση των δημοσιονομικών πόρων, όταν κάθε 6 με 7, 8 μήνες έχετε καινούργιες κυβερνήσεις. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ειλικρινά, τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου, ότι δηλαδή οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην πρόοδο τη νησία στη μετα... περίοδο, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική η διαπίστωση αυτή. Χαίρομαι λοιπόν που και το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και ο εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα και αναγνωρίζουν και την περιπλοκότητα της κατάστασης την οποία πέρασε την Ισία πρόσφατα. Η έκθεση, ας μην το λησμονούμε αυτό, ασχολείται με την περίοδο 2011 έως 2015 και μέγα μέρος της κριτικής που σωστά κάνει ε, το ελεγκτικό συνέδριο έχει στο μεταξύ αντιμετωπιστεί, διότι βρισκόμαστε πλέον στο 2017 και βλέπουμε μια περαιτέρω σταθεροποίηση παρότι που δεν είναι απολύτως εξομαλυμένη κατάσταση, πάντως μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα θέματα που δικαίως φύγουν ελεγκτικό συνέδριο και εισηγητής. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι λοιπόν με την έκθεση, το ξαναλέω, δεχόμαστε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19 ε, ε, η Ιουνίου και την θετική κρίση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 20ης Ιουνίου σχετικά με την αποστολή που διεξήγαγε στην Τινησία πριν ε, από λίγε εβδομάδες και που επέτρεψε στους ευρωβουλευτές να παρατηρήσουν οι ίδιοι επιτόπου και να ειδούν όχι μόνο τις προκλήσεις αλλά και το σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η Τινησία και πώς βοήθησε η δική μας στήριξη. Στην επίσημη πτυχή μπορούμε να επαναλάβουμε την αποδοχή των τεσσάρων συστάσεων του Ελεκτικού συνεδρίου αλλά και των δέκα συστάσεων του εισηγητού σας και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μπορώ να σα πω ότι τα έχουμε γράψει άλλωστε αυτά τα πράγματα, ότι αναμείναμε μέχρι τη σημερινή συζήτηση για να αντιμετωπίσουμε ορισμένε από τι συστάσει που μα έχουν κάνει και το ελεγκτικό συνέδριο και ο εισηγητή. Και ιδίω ο κοινό προγραμματισμό, α μην δυσμονούμε ότι ο κοινό προγραμματισμό έρει τι αρχέ του από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2012 που επαναλήφθηκαν τον Μάιο του 2016 οι υπουργοί κατέστησαν σαφέ ότι ο κοινό προγραμματισμό θα πρέπει να είναι ο κανόνα ταυτόχρονα όμω να είναι οικειοθελές. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων δεν θα πρέπει να αφιστούν προσπαθειών για να προωθήσουν το κοινό πρόγραμμα. Εν τέλει όμω, δεν έχουμε πολιτικά ή άλλα μέσα για να υποχρεώσουμε τι χώρε μέλη να τα εφαρμόσουν τα πράγματα. Αν ξεπεράσουμε λίγο το πλαίσιο τη Τινησία, βλέπουμε διαφορετικά σενάρια. Βλέπουμε χώρε όπου οι χώρε μέλη συμμετέχουν όλε μαζί και θέλουν κοινό προγραμματισμό. Υπάρχουν άλλε περιπτώσει όπου ορισμένε χώρε μέλη θέλουν να συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή σε μια κοινή ανάλυση, άλλο όμω κοινή ανάλυση, άλλο η joint response. Εκεί γίνονται πιο επιλεκτικές. Ορισμένε φορέ δεν θέλουν καθόλου να κινηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Άλλε θέλουν να περιοριστούν σε ορισμένου τομεί, αλλά να αφήσουν άλλου τομεί εκτό του πλαισίου του κοινού προγραμματισμού. Τα λέω αυτά για να σας εξηγήσω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να υλοποιήσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για κάτι το νέο. Από την άποψη αυτή, νομίζω ότι στην περίπτωση της νησίας επιτυγχάνουμε σημαντική πρόοδο, κυρίως όμως τα τελευταία δύο χρόνια. Διότι αποδίδουν τα προγράμματα, υπάρχουν, μηχανισμοί συντονισμού ιδίω μετά το 2015 και σε ορισμένου τομεί θα κάνουμε αυτά. Κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε τώρα στα πλαίσια της διαδικασία να δώσουμε τελική μορφή στο ενιαίο πλαίσιο και στο ε, πλαίσιο γειτονία που αυτά αρχίζουν και γίνονται πραγματικότητα και συνεργαζόμαστε και σε αυτά με τις ε, χώρες μέλη. Έχουμε 18 χώρες μέλη παρούσες στην Τινησία όλες εμπλέκονται στην προσπάθεια αυτή. Έχουμε τώρα το πενταετές σχέδιο αναπτύξεως της Τινησίας, που είναι όχι μόνο κυβερνητική στρατηγική, αλλά την έχει εγκρίνει και το Τινησιακό Κοινοβούλιο. Άρα έχουμε στα χέρια μας τώρα την βάση για το κοινό αυτό πρόγραμμα και προχωρούμε. Πιστεύουμε επίσης ότι έχει δίκιο το ελεγκτικό συνέδριο ότι θα πρέπει να είμαστε πιο στοχευμένοι. Στοχευμένοι και σε ό,τι αφορά την επιλογή των προγραμμάτων που θέλουμε να προωθήσουμε, αλλά και σε ό,τι αφορά του όρου, την αιρεσιμότητα. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τον εκπρόσωπο του Ενεκτικού Συνεδρίου που λέει ότι είμαστε πολύ γενναιόδοροι με την αιρεσιμότητα. Μπορούμε μάλιστα να αποδείξουμε ότι σε ένα αριθμό περιπτώσεων δεν πληρώσαμε τα πάντα που είχαμε υπογράψει να πληρώσουμε, διότι θεωρήσαμε ότι ορισμένοι όροι τη αιρεσιμότητας δεν πληρούνταν. Πρέπει ωστόσο να γίνει διάκριση ανάμεσα σε καθιερωμένες, σε ε, ε, καθορισμένες ε, δόσεις, τις οποίες έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε άμα τη υπογραφή, και άλλες οι οποίες πρέπει να εξαρτηθούν από το ποιοι όροι εκπληρώθηκαν, σε ποιο βαθμό και θα δούμε τότε αν θα πληρώσουμε 100%, 50% ή και 0%. Και αυτό το κάνουμε σε όλες τις χώρες, επομένως και στην Τινησία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν καταβάλαμε το πλήρες ποσό, διότι δεν θεωρήσαμε ότι η αξιολόγησή μας έδινε τη δυνατότητα αυτή. Όσον αφορά τον αριθμό τομέων, είμαι βέβαιος ότι έχει δίκιο το Ελεκτικό συνέδριο ότι πρέπει να περιοριστούμε σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τομέων. Τώρα όμως με τον πεντιετή σχεδιασμό που γνωρίζουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της νησιακής κυβέρνησης έχουμε και μεγαλύτερη σταθερότητα και από πλευράς κοινοβουλίου και από πλευράς της νησιακής κυβέρνησης. Άρα η επιλογή των προτεραιοτήτων τώρα είναι ευκολότερη. Τούτου εκθέτω, ο κ. Σπίνξτεν τα ξέρει άλλωστε αυτά, το ελεγκτικό συνέδριο εξέτασε τι ευρωπαϊκέ ενισχύσει προς την Τινησία σε ένα ευρύτατο φάσμα. Όχι λοιπόν μόνο μικροοικονομική ενίσχυση. Χρησιμοποιούμε 10 και παραπάνω κονδύλια του προϋπολογισμού, σειρές του προϋπολογισμού. Και είναι σαφές ότι όταν χρησιμοποιεί κανείς τέτοιο ευρύ φάσμα γραμμών του προϋπολογισμού, είναι κάπως τεχνητό να πει κανείς ότι πρέπει να περιοριστούμε μοναχά σε τρεις τομείς. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή, αυτό το δεχόμαστε. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υποκείμεθα δεν και καλά σε αυτό το μάντρα του ότι μόνο τρεις τομείς θα πρέπει να είναι αυτοί στους οποίους θα περιοριστούμε. βάζουμε στενότερες στόχους τώρα, ε, κάνουμε και φτιάχνουμε και κλάστερ, ομάδες στόχων. Αυτό θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας των ισχύσεων που θα δίνουμε και μετά το 2015 ήδη με το Single Support Framework που υπάρχει τώρα και που λύγει στα τέλη του έτους έχουμε συγκεκριμένες επιλογές για χρηματοδότηση μικρότερου αριθμού τομέων και κάνουμε και μια αυστηρότερη προσπάθεια τώρα και αυτό μέσα στο πλαίσιο μέχρι το 2020. Επίσης και στις διάφορες ανακοινώσεις που έχουμε συντάξει και στην ανακοίνωση της 29ης Ενάτου πέρσι για την Τινησία και ήταν η πρώτη φορά όπου Επιτροπή, ε, μάλλον, Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων έκαναν μια κοινή ανακοίνωση για μια χώρα. Τώρα για την ε, κριτική ΠΕΦΑ. Συμφωνούμε και εμείς ότι οι πέφα θα πρέπει να οργανώνονται συχνότερα. Χρειαζόμαστε επικαιροποιημένη ΠΕΦΑ. Η συνήθις περίοδος για τις ΠΕΦΑ είναι τέσσερα έτη. Τώρα οφείλουμε να πούμε ωστόσο ότι η πρόσφατη ΠΕΦΑ που, που ε, αναφέρεται στην περίοδο του 2015 εκδόθηκε τούτο τον Απρίλιο, φέτος δηλαδή, και η επόμενη θα είναι σε 2-3 χρόνια. Αυτό έχει σχέση με το γεγονό ότι η μεθοδολογία για τις ΠΕΦΑ έχει αλλάξει. Βεβαίω μα ενδιαφέρει η εξέλιξη αυτή και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πίνξτεν ότι πρόκειται για, σημα... για πολύ σημαντική προπόθεση για την επόμενη δημοσιονομική στήριξη. Τονίζω ακόμη κύριε Πρόεδρε ότι βεβαίω επιμένουμε στο γεγονό ότι η υποστήριξή μα και η πρόοδος αξιολογούνται διαρκώς και για την Τινσία και για άλλες χώρες. Αυτό που δεν έχουμε επί του παρόντος είναι μια συνολική αξιολόγηση χώρας, που δεν το χρειαζόμαστε όμως τώρα, γιατί έχουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Έχουμε όμως αξιολόγηση ανατομέα. Και όσο γνωρίζετε, έχουμε και το σύστημα του Result Oriented Monitoring για κάθε ένα από τα προγράμματα και έργα που μας δίνουν feedback ίσως όχι σε πραγματικό χρόνο, αλλά πάρα πολύ σύντομα μετά από την ε, απόδοση του προγράμματος και μπορούμε να εξασφαλίσουμε ώστε η αξιολόγηση να είναι ρεαλιστική, εγγύς και να μας δίνει τις δυνατότητες προσαρμογής των προγραμμάτων όταν βλέπουμε τη σχετική ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, not too much. Ναι. Νομίζω πως δεν υπάρχουν πολλά στα οποία χρειάζεται να απαντήσετε μόνο ένα-δυο σχόλια, οπότε ας ακούσουμε τα τελικά σχόλια. Ναι, Πρόεδρε, ένα μόνο σχόλιο θα κάνω. Ένα μόνο ζήτημα θα θέξω. Για να είμαι κι εγώ στοχευμένος. Σε ό,τι αφορά ε, την ε, διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε, δηλαδή Επιτροπή, μέλος εδώ της Επιτροπής και Ελεκτικό Συνέδριο. Η χρηστή οικονομική λοιπόν δημοσιονομική διαχείριση είναι πάρα πολύ σημαντική όταν, υπάρχει, όταν βλέπονται κονδύλια τα οποία δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω πως θα πρέπει να συμφωνήσει η Επιτροπή. Εάν δούμε για παράδειγμα το ΠΕΦΑ 2015 που το έχω μπροστά μου, ποια είναι το rating, ποιο, η αξιολόγηση δηλαδή, η βαθμολογία BC. Δηλαδή το πρώτο τελευταίο αν θέλετε κατόφληση σε διεθνές επίπεδο. Άρα κάτι θα πρέπει να γίνει στο επίπεδο της χρηστής νοσομικής διαχείρισης από πλευρά της Τινησίας. Ε, νομίζω ως προς τα υπόλοιπα συμφωνούμε μεταξύ μας για τα γενικά συμπεράσματα. Είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε, είναι θετικά, υπάρχουν κάποια σημεία επιμέρους ε, κριτικής, αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να επιλύσουμε είναι το ζήτημα της χρηστής νοσομικής διαχείρισης. Ο κ. Σπανό. Απλώς και πάλι να ευχαριστήσω το αλλά βέβαια και να ευχαριστήσω για την εργασία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την ποιότητα των απαντήσεων που δόθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι οι συστάσεις του λεπτικού συνεδρίου αυτά που είπε ο κ. Πίξτεν συμπίπτουν αυτά τα οποία εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών ε, παρέχουμε. Γιατί είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Ούτω ώστε η χώρα η συνεχίζει και βρίσκεται σε δυσκολίε, ε, συμβάλλουν λίγο αυτέ οι συστάσει για να υπερκυράσει τι δυσκολίε η χώρα. Και πρέπει επομένω ε, προ το συμφέρον τη χώρα αλλά και προ το συμφέρον ημών των Ευρωπαίων να προσπαθήσει η χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ολοκληρωμένη αυτή η συζήτηση και χαίρομαι που συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Άρα, ωραία. Διάφορα ενεχματίποτε, προσεχή συνεδριάσεις, 12 Ιουλίου, 17 είναι η επόμενη συνάντηση, πέρα συνεδριάσεις. Ευχαριστώ.